Καλό σας απόγευμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω την κυρία Σαμπίν ε, Λαριουέλ, ε, Βελγίδα Υπουργό Γεωργίας και επομένως Προεδρεύουσα ε, του Συμβουλίου είναι εκπρόσωπο επομένω τη απερχόμενη Προεδρία. Εγκρίνουμε λοιπόν την ημερησία διάταξη, και δεν υπάρχουν σχόλια και παρατηρήσει. Να εγκρίνουμε επίση και τα πρακτικά των συνεδρίων τη 15η Νοεμβρίου, 18η Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου 2010. Εάν δεν υπάρχουν ε, σχόλια μέχρι το τέλο τη σημερινή συνεδρίασης, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Να σας κοινοποιήσω επίσης ότι έχουμε web streaming αυτής της ε, συνεδρίασης. Και, ε, Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Σαμπίν ε, Λαριουέλ. Αγαπητή Σαμπίν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εργασία την ε, οποία ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια της καρποφόρας, του καρποφόρου συγγνώμη, εξαμήνου έχεις κάνει και σου δίνω τον λόγο λοιπόν σαν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Γεωργίας. Σαμπίν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η Βελγική Προεδρία, όπως γνωρίζετε όλοι, ολοκληρώθηκε τέλη Δεκεμβρίου ε, και νομίζω ότι καταφέραμε να προχωρήσουμε σε κάποια θέματα. Βεβαίως, δεν θα σας υπενθυμίσω ότι η Βελγική Προεδρία εγγράφεται ε, στα πλαίσια μιας προεδρίας ε, σε τρία σκέλη, ε, δηλαδή συνεργασία με την απερχόμενη Ισπανική Προεδρία, ε, την δικιά μας και την επόμενη τωρινή πλέον Ουγγρική Προεδρία. Επίσης η Βελγική Προεδρία ε, ξεκίνησε κάποια ειδική στιγμή, όπου δηλαδή είχε ξεκινήσει η συναπόφαση βάσει της νέας συνθήκης της Λισαβόνας και που έδωσε νέες εξουσίες στο Κοινοβούλιο και βεβαίως εδώ να ευχαριστήσω τον αγαπητό Παόλο για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών. Ε, θα σας παρουσιάσω κάποια, κάποιους φακέλους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ξέρω ότι επισταμένως εργάζεστε επί του θέματος αυτού και βεβαίως είναι ένα ζήτημα ε, στο οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε κάποια στιγμή, αλλά που εν πάση περιπτώσει προσπάθησε η Βελική Προεδρία ε, να το προετοιμάσει, να προετοιμάσει τις συζητήσεις, να προετοιμάσει επίσης και την εργασία που έκανε η Επιτροπή δια του αντιστοίχου αρμοδίου καθήλυνα Επιτρόπου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στην ΛΑΙΛΠ και την παρουσία μάλιστα του Προέδρου, ε, την παρουσία του Πάολο, ε, συζητήσαμε κάποια θέματα επί των οποίων είχαμε την δυνατότητα σε μεγάλη πλειοψηφία στα πλαίσια των 27 χωρών μελών να θίξουμε κάποια ε, θέματα υπενθυμίσαμε την επιθυμία μας, ε, κάτι που μπορεί να φαίνεται αυτονόητο όταν μιλάμε μεταξύ Υπουργών ε, Γεωργίας, αλλά είναι καλό να το τονίζουμε ε, προς όλα τα ότα ε, ότι δηλαδή επιθυμούμε μια ισχυρή και πραγματικά κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης είπαμε ότι θέλουμε αυτή την ΚΑΠ η οποία θα φασίζεται σε δύο πυλώνες. Ε, έναν πυλώνα που θα ελέγχεται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αφορά τα μέτρα ε, για την αγορά και τα μέτρα της διατροφικής ασφάλειας καθώς επίσης και θέματα όπως είναι χωροταξικά, χωροταξικές αλλαγές, κλιματικές αλλαγές και ένα δεύτερο πυλώνα που κατά την άποψή μα θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο και η κατανομή μεταξύ των δύο πυλώνων, αυτό είπαμε και το Σεπτέμβριο στην ΑΕΛΠ, μα ε, φαίνεται ότι θα πρέπει να είναι καλύτερα αποσαφινισμένο έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, διάβια εξαφήνεια μεταξύ των, ε, των δύο πυλώνων. Ε, αλλά και από την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στι απαιτήσει του δευτέρου πυλώνα που βεβαίω θα, ε, εμπίπτει στην συγχρηματοδότηση. Ε, ε, ε μεγάλη αλλαγή τιμών, την ποιοτικότητα της αγοράς, την, τις μεγάλες διακυμάνσεις τιμών. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και υπενθυμίσαμε ότι η ενισχυμένη, μεταρρυθμισμένη κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να δώσει την δυνατότητα να ανταποκριθούμε καλύτερα στα προβλήματα αυτά και βεβαίως να δώσουμε καλύτερες δυνατότητες, δηλαδή θέλω να πω ε, να υφίστανται οι γεωργοί το εισόδημά τους μικρότερες διακοιμάνσεις. Δεν λέω ότι θα πρέπει μία φορά ε, ε, να καθορίσουμε τον μισθό, της απολαβές των γεωργών, αλλά βεβαίως για να διατηρήσουμε την ζωτικότητα ε, της ε, υπαίθρου θα πρέπει ε, να έχουν και κάποια, κάποια σταθερότητα οι γεωργοί και επομένως θα πρέπει να μειωθεί η υπερβολική συγκυριακή διακύμηση των τιμών. Επίσης δώσαμε δυνατότητα στον ε, Επίτροπο κάποιες ιδέες έτσι ώστε ε, να ε, κάνει τις ανακοινώσεις του. Τον Νοέμβριο στο Συμβούλιο ακούσαμε τις απόψεις ε, είπαμε ότι σε γενικές γραμμές και επί των ε, κυριωτέρων αρχών υπήρχε μάλλον ομοφωνία και μετά αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία ε, συζήτηση σχετικά με το πρώτο θέμα που όρισε ο, ο, Επίτροπος, δηλαδή στις 13 Δεκεμβρίου είχαμε αποφασίσει να συζητήσουμε για την ανταγωνιστικότητα και για την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η Ουγγρική Προεδρία. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι και εσείς θα μπορούσατε ίσως να δουλέψετε πάνω στο θέμα αυτό έτσι ώστε ε, να ε, αντιμετωπίσουμε από κοινού όλα τα θέματα. Εμείς οργανώσαμε και, μία, και ένα γεύμα εργασίας ε, πάνω σε αυτήν την ιδέα της ενεργητικής γεωργίας. Για την ώρα σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, αναγνωρίζουν ότι αυτή η ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά βεβαίως ε, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, έτσι δεν είναι τόσο απλοϊκά. Πάντως είχαμε μια καλή πρώτη ανταλλαγή απόψε. Δεύτερο φάκελος, ε, πάρα πολύ σημαντικός, ο φάκελος του γάλακτος. Όχι ομόφωνα, αλλά κατά 75% υπερψηφίστηκαν τα συμπεράσματα στο Συμβούλιο της 27ης Σεπτεμβρίου και η Βελγική Προεδρία ήταν της άποψης ότι θα έπρεπε να δουλέψει κυρίως επί της ουσίας, δηλαδή όχι να γίνουν απλώς συμπεράσματα κενά νοήματος ε, τα οποία όμως θα ετύχαναν του 100% της ε, ε, συμφωνίας. Η Βελική Προεδρία λοιπόν επέλεξε την οδό της δυσκολίας, επομένως πιο δύσκολη ουσία, άρα 75% πλειοψηφίας. Επίσης, συζητήσαμε την 13η Δεκεμβρίου για τις προτάσεις και την έκβαση της ε, υψηλού επίπεδου ομάδας ε, για το γάλα. Ξέρετε, όπως και εγώ άλλωστε, ότι γίνονται πολλές συζητήσεις τώρα. Αυτή η ιδέα της σύμβασης είναι πολύ υποσυζήτηση. Τι θα γίνει έτσι ή αλλιώς ε, θα δούμε. Θα δούμε Νομίζω ότι όλοι πάντως συμφωνούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε περαιτέρω, ε, να συνεχίσουμε και οπωσδήποτε οι γεωργοί να έχουν μεγαλύτερο διαπραγματευτικό βάρος. Τρίτη δέσμη, τρίτος φάκελος είναι το, ο φάκελος της ποιότητας που μας απασχόλησε στην Προεδρία. Δυστυχώς τα κείμενα της Επιτροπής μας έφτασαν μόλις την 10η Δεκεμβρίου έχοντας οργανώσει το Συμβούλιο για την 13η Δεκεμβρίου. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες αλλά η ποιότητα είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα και η πρόταση ε, κανονισμού για τον ποιοτικό έλεγχο ε, των ε, γεωργικών προϊόντων θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα στο ευρύτερο και συνολικό πρόγραμμα ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω διαπραγματεύσεις λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξουν επιμέρους τομεακοί κανονισμοί και βεβαίως νέες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για το προαιρετικό πρόγραμμα ελέγχου ε, στην ε, σήμανση των προϊόντων. Ε, και βεβαίως αυτό θα ενσωματωθεί και με το προηγούμενο ζήτημα του γάλακτος. Κάναμε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων και δώσαμε τη σκητάλη τώρα στην Ουγγρική Προεδρία. Τέταρτο ζήτημα, τέταρτος φάκελο. σημαντικό για όλη την και για το Βέλγιο αλλά και για την ε, κτηνοτροφία το ζήτημα της πονκόδου συγκεφαλοπάθειας ε, και στο ε, ζήτημα αυτό είχαμε την δυνατότητα την 29η Νοεμβρίου να εγκρίνουμε ομόφωνα αυτή τη φορά κάποια τα συμπεράσματα κυρίως στα σημεία στα οποία είχαν καταλήξει οι εμπειρογνώμονες στους οποίους είχαμε ζητήσει μελέτες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 πέμπτο σημείο ε, όπου κυρίως ενδιαφέρει τη Γερμανία, είναι γερμανικό το μονοπόλιο αλλά είναι η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνης είναι, ε, ε, και βεβαίως όταν κάνουμε απολογισμό υπάρχουν θετικά στοιχεία κύριε Πρόεδρε τα οποία μας ικανοποιούν αυτά που σας ανέφερα μέχρι τώρα αλλά υπάρχουν δυστυχώς και ζητήματα επί των οποίων θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε κάπου. Το πρώτο λοιπόν ε, θέμα ε, είναι το ζήτημα που αφορά τους ε, γενετικώς τροποποιημένους με οργανισμούς. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ επιφυλακτική η υποδοχή του κειμένου και το επιφυλακτικό, ε, επιφυλακτική είναι ένα πολύ διπλωματικό επίθετο το οποίο χρησιμοποιώ. Ε, οπότε κουμποθήκαμε, δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Και τελευταίος φάκελος που θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο, δεν καταλήξαμε όμως πουθενά και αποφάσισα τελικά να μην το εγγράψω εις ε, το Συμβούλιο του Νοεμβρίου γιατί υπήρχε ανασχετική πλειοψηφία η οποία Διαρκώ διαρκώς απέριπτε το θέμα ήταν η βοήθεια προς τους πλέον ενδεείς Προσπαθήσαμε λίγο να ξεμπλοκάρουμε το θέμα, αλλά ούτως ή άλλως ε, ε, διεφαίνεται η κατάσταση ότι θα οδηγηθεί δηλαδή σε μια ανασχετική πλειοψηφία, ε, συγγνώμη, ανασχετική μειοψηφία και επομένως προσπαθήσαμε να μιλήσουμε κυρίως με το Κοινοβούλιο, με τον Επίτροπο Νταλή έτσι ώστε να επανέλθει λίγο στις προτάσεις όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση, αλλά ε, βάσει συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας, την οποία μπορώ να κατανοήσω φυσικά, ε, δεν θέλησε να προχωρήσουμε περισσότερο ε, στην συζήτηση αυτή. Πιστεύω ότι είναι λυπηρό που δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε αυτό το θέμα ε, για τους ε, έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη και το Βέλγιο και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα βοηθούσε πολύ την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτά ήθελα να σας πω εν είδη γενικής ε, έποψης ε, κύριε Πρόεδρε, μια γενική παρουσίαση και βεβαίως εξ αρχής σας λέω ότι είμαι στη διάθεσή σας με μεγάλη χαρά να απαντήσω σε σχόλια, ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ Σαμπίν, λέει ο Πρόεδρος, και σε ευχαριστώ και για την ουσία και για το περιεχόμενο της εργασίας σου και για τον τρόπο με τον οποίο μας παρουσίασες το εξάμεινο της Βελγικής Προεδρίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους αγορητές. Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε το λόγο ως ήθιστε ή στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά θα ε, συνεχίσουμε. Συντονιστής λοιπόν του ΕΛΚ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό για την ε, παρουσίαση των τεκτενωμένων της Βελγικής Προεδρίας και αναφερθήκατε σε μία σειρά από θέματα τα οποία επεξεργαστήκατε κατά την θητεία σας και θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ήταν εύκολη κατάσταση και γι' αυτό είναι σωστό να επενέσουμε το ότι εσείς ε, ε, σημειώσατε τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Αναφερθήκατε στην αναθεώρηση της γεωργικής πολιτικής και αιτιολογήσατε γιατί χρειαζόμαστε αυτή την κοινή γεωργική προεκλητική, ιδίω για τη διατροφική ασφάλεια και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί ομιλούμε διότι είπατε ότι πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή γεωργική πολιτική το σαν κοινοβούλιο χρειαζόμαστε το Συμβούλιο για να μπορέσει να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση για την κατάλληλη γεωργική πολιτική και όσον αφορά τον διαχωρισμό του πρώτου και του δευτέρου πυλώνα τον οποίον ζητήσατε είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μια, ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ της πρώτης και του πρώτου και του δευτέρου πυλώνα και ο δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να διαμορφωθεί πιο ευέλικτα. Είμαι εισηγητής για αυτή την αναθεώρηση της γεωργίας και διεξάγω αυτή την εποχή πολλές συζητήσεις. Ασχολούμαι 10 χρόνια με τη γεωργική πολιτική και βλέπω τώρα που υπάρχουν συζητήσεις με 27 κράτη-μέλη πόσο διαφορετική και επιπυλόμορφη είναι η Ευρώπη και θα συνεχίσει είναι και γι' αυτό θα χρειαστούμε και στο μέλλον ευελιξία. Δεν χρειαζόμαστε ε, μία πολιτική η οποία από τις Βρυξέλλες θα προδιαγράφει τι θα γίνεται στα 27 κράτη. Γι' αυτό και θα ήθελα να κάνετε λίγα περισσότερα σχόλια για το ότι θα επιθυμούσατε να λάβουμε υπόψη από βελγικής απόψεως εις ε, τον δεύτερο πυλώνα διότι έτσι μπορεί να υπάρξουν θέματα τα οποία θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας και επίσης δεν θέλω να υφαρπάξω τον χρόνο των συναδέλφων παρόλο που θα είχα πολλά να πω ακόμη αλλά υπάρχουν διακοιμάσεις των γεωργικών τιμών και ε, ε, δεδομένης της καταστάσεως ε, ίσως μπορείτε να μας προτείνετε πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτές τις διακυμάνσεις διότι θυμάμαι ότι ο Γάλλος ο πρόεδρος Σαρκοζή είχε στην εποχή του εκφραστεί πολύ σαφώς ότι πρέπει να ε, να χρησιμοποιήσουμε ε, όλες τις, ε, όλα τα θέματα τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στην έκθεση την οποία καταρτίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο συντονιστής τώρα των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας συγχαρώ για την καταπληκτική δουλειά σας και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην προσωπική σας ζωή και στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, εγχώρια προβλήματα στο Βέλγιο και ελπίζουμε να υπερπηδηθούν το στομότερο δυνατό. Πάντως το Βέλγιο ε, ήταν πάρα πολύ ικανό ε, στην άσκηση της Προεδρίας και αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Παρά τα προβλήματα που έχουμε βιώσει τους τελευταίους έξι μήνες και συγκεκριμένα και στον τομέα της γεωργίας, Ξέρουμε ότι ήταν ένα επιτυχημένο εξάμεινο σε σχέση με την ε, διαχείριση και της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής. Η Επιτροπή έχει κάνει κάποια συμπεράσματα για το γαλακτοκομικό τομέα, για τον τομέα του γάλακτος, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ευφιές το ξεκίνημα της Βελγικής Προεδρίας ε, σε ό,τι αφορά την δρομολόγηση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Έτσι έχουμε πλέον καλές προοπτικές για ευόδοση των διαπραγματεύσεων και βασίζομαι και ε, στις ικανότητες του συναδέλφου Ντές, θα συζητήσουμε μαζί ε, το θέμα αυτό. Είναι το κλειδί της μελλοντική γεωργίας. Είμαστε σε μεταβαλλόμενους καιρούς και θα πρέπει να μπορούμε την πολιτική αυτή που αποτελεί τμήμα της ιστορίας μας να την μεταλαμπαδεύσουμε και στους μελλοντικού ε, Ευρωπαίους πολίτες και στις μελλοντικέ γενιές. Και θέλουμε βέβαια αργότερα να συζητήσουμε και με τον Ούγκρο ομολογό σας κάποια από αυτά που αναφέρατε εσείς. Πάντως εσείς τα πήγατε περίφημα. Τα πήγατε καταπληκτικά και εκ μέρους πολιτικής μου ομάδας, αλλά φαντάζομαι και όλων των άλλων ε, σας Ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον. Ευχαριστώ, Λουίς. Ο Γιώ Λάινεν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την βελγική κυβέρνηση για την εξαιρετική εξάμεινη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία ήταν πάντα σταθερή και έγινε, προσ... έγινε πρόοδος σε αρκετά ε, ζητήματα. Και βεβαίω ε, όσον αφορά την μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής είχαμε την ανακοίνωση της Επιτροπής και φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία στην, στο παρόν Συμβούλιο Γεωργίας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Τώρα, Ε, θα ήθελα να μας πείτε αν ε, έχετε την αίσθηση ότι το Συμβούλιο θέλει πραγματικά μια κανονική μεταρρύθμιση ή αν θέλει κάποιες μικρές αλλαγές που όμως ε, θα επιτρέψουν στην, στο status quo να διατηρηθεί. Ε, μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε στην, ε, στο, στη, στη νέα περίοδο 13-20 ε, και βεβαίως θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να μεταστρέψουμε την στρατηγική μας, την πολιτική μας έτσι ώστε να είναι πιο στοχευμένη. Επίσης, όσον αφορά την ανταγωνιστική γεωργία αλλά και την αηφόρο γεωργία. Ε, μερικοί έχουν την εντύπωση ότι αυτά τα δύο θέματα είναι, ε, βρίσκονται σε αντιπαράθεση, είναι ε, αντικρουόμενα μεταξύ τους. Εγώ δεν το πιστεύω. Θα ήθελα όμως την άποψή σας σχετικά με τους δύο αυτούς στόχους που θα πρέπει να επιδιώξουμε στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την τεράστια αύξηση κατά 50% των ε, διατροφικών ε, απαιτήσεων της ζήτησης σε διατροφικά ε, είδη μια και αυξάνεται και ο πληθυσμός του πλανήτη. Θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας επίσης ε, για μια πιο ανταγωνιστική γεωργία ή προς μια αηφόρο γεωργία. Θεωρείτε ότι είναι ένας διτός στόχος τον οποίο μπορούμε ε, να επιτύχουμε από κοινού ή, ε, ή τον έναν ή τον άλλον. Κυρία Υπουργό, Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ όπως και οι συνάδελφοι για την διεξαγωγή της προεδρίας σας. είμαστε τυχεροί γιατί η μεγάλη κρίση του γάλακτος ε, στο τέλος του έτους ε, ε, μπόρεσε να ηρεμήσει και ανέβηκαν λίγο οι τιμές. Θα, θα επανέλθω στο θέμα του γάλατος γιατί ε, η, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δίνει ε, μεγαλύτερες δυνατότητες στους παραγωγούς ε, να συσπηρωθούν δεν είναι ε, φιλόδοξη δεν υπήρξε αρκετό θάρρος θα έλεγα ιδίως σε αυτό το τομέα και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου να πούμε ότι οι αγορές πρέπει να ρυθμιστούν, οι γεωργοί πρέπει να μπορούν να οργανωθούν και όπως άλλωστε είπαμε πρέπει να δώσουμε ένα μεγαλύτερο μέρος της διατροφικής αγοράς ή στους γεωργούς, πράγμα το οποίο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής η ανακοίνωση πέρυσι ε, ξένησε πολλούς, διότι ουσιαστικά δεν είχε τη μορφή που πολλοί ανέμεναν. Δηλαδή δεν ήταν πολύ συγκεκριμένοι σε πολλά θέματα και ίσως είναι καλό αυτό διότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τώρα τη δυνατότητα να κάνουμε μία κοινή συζήτηση και ε, να καθορίσουμε ένα πλαίσιο, να γεμίσουμε το πλαίσιο το οποίο έχει ε, να φέρει μόνο επιγραμματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνδυάσουμε την γεωργική πολιτική με τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι γιατί από τη μία πλευρά πρέπει να αναθεωρήσουμε χωρίς να ξέρουμε τι δημοσιονομικές δυνατότητες θα υπάρξουν και στο τέλος τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την κοινή γεωργική πολιτική. Ακούσαμε πολλούς επένους για την κοινή γεωργική πολιτική από πολλά κράτη αλλά ξέρουμε ότι πολλά κράτη στην ε, ε, ουσία ε, προβαίνουν σε και ε, πρέπει να ξέρουμε τι επιδιώκουμε με τη γεωργική πολιτική και αν θέλουμε μία αναθεώρηση της γεωργικής πολιτικής πρέπει να τη χρηματοδοτήσουμε κιόλας. Ε, πέραν αυτού πρέπει να συνεργαστούμε. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν το θέμα της διατροφικής ασφάλειας που θα είναι πολύ σημαντικό τα επόμενα έτη για να ξέρουμε τι δημιούργησε και θα δημιουργεί και στο μέλλον της κρίσης, δηλαδή η κερδοσκοπία. Η κερδοσκοπία προκάλεσε ε, την ε, κρίση των τροφίμων και πρέπει από κοινού, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και από άλλες πλευρές να θέσουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο, διότι ξέρω ότι ο Γάλλος Πρόεδρος έχει θέσει ένα ενδιαφέρον πλαίσιο, αλλά θα πρέπει ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε περισσότερα πράγματα από κοινού, διότι ε, ουσιαστικά αυτό που μας απασχολεί δεν είναι ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά διεθνές και επίσης μιλήσατε για την επανεθνικοποίηση της γενετικής πολιτικής. Ίσως θα μου εξηγήσετε ποια είναι η θέση του, της πλειοψηφίας του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή διότι αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι εάν τα κράτη θα διατηρήσουν το δικαίωμα της αδειοδότησης και επίσης ε, κατά πόσο ε, μια κοινή αγορά μπορεί ε, να συμβιβάζεται με μια επανεθνικοποίηση της αδειοδοτήσεως και να δούμε πού υπάρχουν κοινά σημεία, δηλαδή πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τους επόμενους μήνες. Ε, θέσατε πολλά ενδιαφέροντα ενάυσματα, ε, πολλά θέματα ε, δεν απο δεν τα αποκρύψατε και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα μπορέσουμε να τα συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ Μάρτιν. Ο Λορέντσο Φοντάνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Υπουργό για την παρουσία της εδώ. Την ε, συγχαίρω και εγώ για αυτό το ε, εξάμεινο της Βελικής Προεδρίας που δούλεψε τόσο πολύ καλά. Απόψή μας ε, είναι ότι βεβαίως χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα είναι επικεντρωμένη στην ποιότητα, άλλωστε έγινε και έκθεση για το θέμα αυτό και να δούμε πώς στο εγγύς μέλλον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της σήμανσης των ετικετών αλλά θα θέλαμε και την άποψή σας σχετικά με τις εισαγωγές στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, φαντάζομαι, συχνά ε, γίνονται εισαγωγές οι οποίες βεβαίως δεν, δεν σέβονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άρα οδηγούν ε, σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Υπάρχουν και κάποιοι ε, πολύ ισχυρές παράμετροι, κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν για το μέλλον. Και θα θέλαμε μια γενικότερη αξιολόγηση από την πλευρά σας. Ευχαριστώ Λορέντζο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ε, ο κύκλος των ε, συντονιστών. Από την Κούε τώρα ο κύριος Ρούμπι. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους που έλαβαν ήδη το λόγο πριν από εμένα. Και θα ήθελα και εγώ να αναγνωρίσω την ποιότητα του έργου της Βελγικής Προεδρίας στον τομέα της γεωργίας. Έχουμε αφήσει πίσω μας λοιπόν σκληρή δουλειά. Είχαμε μια δύσκολη χρονιά με δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, φυσικά τη δημοσιονομική κρίση. Δεν πέρασε και η Γεωργία Βρόξη Ποσία από όλη αυτή τη διαδικασία. Η Βελγική Προεδρία νομίζω από αυτές τις συνθήκες εξασφάλισε ότι μπορούμε από κοινού να προστατεύσουμε το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Η Ευρώπη έχει αν θέλετε να τακτήσει το σήμα ποιότητας, έχουμε τους δύο πυλώνες, αλλά θα πρέπει να είναι περισσότερο δημοκρατική και περισσότερο υπεύθυνη σε σχέση με το τι μπορούν και το τι δεν μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Εδώ υπάρχει ένα θέμα δύσκολο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και συγκεκριμένα μιλάω για την τιμή, τις τιμές των, αγρο... των γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να εξετάσουμε, να μελετήσουμε την αγορά, την αλυσίδα διανομής. Πολλά κομμάτια αυτής της αλυσίδας ε, ενεργούν ε, με κερδοσκοπικό τρόπο και έτσι πιέζουν προς τα πάνω τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Αυτό νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να το δούμε. Στη Λετωνία, για παράδειγμα, πρόσφατα, οι τιμές των γεωργικών προϊόντων ανέβηκε κατά 20 με 30%. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με τη δική σας προσέγγιση. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Τρόικας, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και με τις άμεσες πληρωμές. Αυτά θα ήθελα. Αλλά σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως για την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ξαναδώσω αμέσως το λόγο στην ε, Υπουργό κυρία Σαμπίν ε, Λαριουέλ έτσι ώστε να απαντήσει στις ερωτήσεις των συντονιστών και μετά θα συνεχίσουμε. Σαμπίν. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αναθέμα και όχι αναβουλευτή. Ε, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους για τις παροτρύνσεις προς το πρόσωπό μου και σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να συνεργαζόμαστε βέβαια και με το Κοινοβούλιο αλλά και με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάντως για τα καλά σας λόγια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία στα οποία αναφερθήκατε. Πρώτα απ' όλα, κοινή γεωργική πολιτική. Μου λέτε κάποιοι πρώτα μήπως πρέπει να περιμένουμε τον προπολογισμό και μετά να δούμε τι γίνεται με την ΚΑΠ. Κοιτάξτε, αν είχα επιλέξει αυτή την επιλογή σήμερα θα μου λέγατε το αντίστροφο. Όλοι ξέρουμε ότι χρειάζεται η κότα και χρειάζεται και το αυγό. Ποιο ήρθε πρώτο δεν το ξέρουμε, αλλά χρειάζονται και τα δύο. Γεωργία, για τη Γεωργία μιλάμε τώρα. Αν λοιπόν περιμένουμε τον προπολογισμό και μετά να καθορίσουμε του μεγάλου στόχου τη κοινή γεωργική πολιτική, θα δώσουμε επιχειρήματα σε αυτού οι οποίοι δεν επιθυμούν πλέον να υπάρχει μια φιλόδοξη κάπ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι. Δίνουμε επίση επιχειρήματα σε κάποιους ηθήνοντες ε, των κυβερνήσεων. Δεν ε, θέλω να πω κάποιον, κατονομάσω κάποιον. Απλά κάποιοι λένε ότι ε, πρέπει να δώσουμε για την ΚΑΠ, πρέπει να δώσουμε για την έρευνα, πρέπει να δώσουμε για την εκπαίδευση κτλ. Άρα εμείς κάναμε μια επιλογή, είπαμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και θα είμαστε όλοι μαζί, οι Υπουργοί Γεωργίας, η Κομισιόν, ελπίζω, πολύ πιο ισχυροί όταν θα πάμε στους υπεύθυνου οικονομικών των κυβερνήσεων και να τους πούμε ότι θέλουμε μια φιλόδοξη ΚΑΠ, άρα πρέπει και ο προπλογισμός να είναι φιλόδοξος. Εγώ δεν είμαι ούτε από αυτούς, ούτε από αυτές συγκεκριμένα που λένε ότι η ΚΑΠ είναι το 40% του προπολογισμού και η έρευνα είναι πολύ Λιγότεροι όσον αφορά το ποσοστό. Είναι λάθος αυτή η συλλογιστική. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τις πολιτικές ε, πλέον στην, ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να κοιτάμε και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό αλλά και τους εθνικούς προπολογισμούς. Γιατί αυτό που έχει γίνει στην Γεωργία είναι ότι λέμε δεν κάνει ο καθένα μόνο του την πολιτική του χωριστά, αλλά προσφέρουμε τα μέσα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Και αν αύριο 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάνουν τι επιλογέ του και ορίσουν το προπολισμό, θα δούμε ε, πώ θα προχωρήσουμε. Όταν κάνουμε λοιπόν συγκρίσει, πρέπει να κάνουμε σωστέ συγκρίσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάπουλα Σάντος που είπε για τη μελλοντική μου πολιτική σταδρομή και για το πολιτικό μέλλον στη χώρα μου που είναι λίγο σκοτεινό προς το παρόν, δεν ξέρουμε προς τα που οδεύουμε και σε σχέση με την κατάσταση του προπολογισμού που πρέπει να έχουμε για να σεβαστούμε αυτά που έχουν αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ πάντως προσωπικά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την κοινή γεωργική πολιτική ως πολιτικός στο Βέλγιο και βέβαια θα αγωνιστώ και για να έχουμε την κατάλληλη την επαρκή χρηματοδότηση για να έχουμε ποιοτική διατροφή, διαφοροποιημένη, ε, να έχουμε ποσότητα, να έχουμε αγρότες. Ε, για όλα αυτά χρειάζονται πόροι. Αν δεν υπάρχουν πόροι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Ο κύριος Λάιον με ρώτησε πριν αν ε, ο στόχος ανταγωνιστικότητα, προμηθευτές τροφίμων και βιώσιμων να πως εκεί υπάρχει κάποια αναντιστοιχία σε ό,τι αφορά την αηφόρα ανάπτυξη, ε, θυμάμαι ότι είναι τρει στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από κοινού. Οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο. Και η Ευρωπαϊκή Γεωργία, η κοινή γεωργική πολιτική, φυσικά και θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτού του τρει άξονε, αυτού του τρει στόχου. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Αλλά πραγματικά είμαι πεπισμένη ότι αν δεν τα καταφέρουμε, είτε από τη μια οι γεωργοί δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκόσμιας διατροφής, της αλλαγής του κλίματος, είτε, να φετέρου θα ε, ανακολουθήσουμε την οικονομική κατεύθυνση και όχι το περιβάλλον και την εφορανέκουση, τότε δεν θα μπορεί να, το, και το κοινωνικό μάλλον, δεν θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους πολίτες αυτά που χρειάζονται. Ο κύριος Λάιον βλέπω ότι δεν είναι ακόμη μέσα, αλλά θέλω να πω ότι το Συμβούλιο Γεωργίας γνωρίζει ότι θα απαιτηθεί μεταρρύθμιση, που θα πρέπει να είναι φιλόδοξη. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο στο Συμβούλιο των 27. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο όραμα, αλλά αυτό που έχουμε κοινό είναι ότι ξέρουμε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση, χρειάζονται προϋπολογισμοί. Και θέλω να σας πω ότι εκεί για τον προπολογισμό κάποιοι θέλουν να μειωθεί ο γεωρικός προπολογισμό και κάποιοι θέλουν να αυξηθεί. Δεν υπάρχει συνένεση ακόμη. Θέλουμε να έχουμε τις δύο πυλώνες, συγχρηματοδότηση και χρηματοδότηση 100%. Από αυτού υπάρχει συμφωνία, όχι όμως σε καμία περίπτωση μάλιστα σε ό,τι αφορά την ισορροπία, την αναλογία. Κάποιοι θέλουν 50-50, κάποιοι θέλουν 80-20 και ίσως κάποιοι θέλουν το 20-80. Άρα δεν έχουμε ακόμη κοινή θέση. Αυτό το οποίο επιθυμούμε να γίνει σε επίπεδο Συμβουλίου Γεωργίας είναι αυτό το οποίο πάντοτε κάναμε στο Συμβουλίο Υπουργών Γεωργίας, δηλαδή να καταλήξουμε, να καταλήξουμε με μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση που τελικά όλοι θα ε, την θεωρήσουν θετική, που δεν θα είναι κάτι εύκολο βέβαια. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε την απαραίτητη ευελιξία στην πτυχή, στην εδαφική και την ιδιαιτερότητα. Ο κύριος Δέσμου είπε τι πιστεύετε για αυτό το δεύτερο πυλώνα. Κοιτάξτε, περιβαλλοντικά μέτρα πιο φιλόδοξα από αυτά που απαιτούνται στον πρώτο πυλώνα. Έχουμε την αρχή των προϋποθέσεων, το conditionality. Θα δούμε και με, τη, με τον πρώτο πυλώνα τι θα συμπεριληφθεί. Σίγουρα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τις αμοιβέ στο δεύτερο πυλώνα. Εκπαίδευση επίσης, καινοτομία το συζητήσαμε χθες στο Συμβούλιο Γεωργίας. Αλλά θέλουμε να ενταχθεί η καινοτομία στις γεωργικές πρακτικές. Άρα χρειάζεται μεταφορά τεχνογνωσίας, χρειάζεται εκπαίδευση, κατάρτιση, επενδύσεις βέβαια και επίσης δυνατότητα να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν σε κάποιες ιδιαιτερότητες ή σε κάποιες συμφορήσεις, προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν ή εδαφικά, ε, ιδιαιτερότητες. Ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις και τη μεταβλητότητα, ναι, πράγματι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο μέτρο παντού. Συμφωνώ, ε, το είπε και η Γαλλική Προεδρία του G20 και ο Γάλλος Νάλφος είπε χθες ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη συνεδρίαση στο πλαίσιο του G20 για την γεωργία. Για το θέμα αυτό ακριβώς, της μεταβλητότητας των διακυμάνσεων. Τι μιλάμε για τον πληθωρισμό, ο Ντάτσιαν Τσιόλος ε, έχει κάνει και αυτό στις δικές του σκέψεις, ε, ο Επίτροπος, το πώς μπορούμε να μειώσουμε την κερδοσκοπία για τις γεωργικέ πρωτεσίλες, αν χρειάζονται ή όχι στρατηγικά αποθέματα και αν ναι, πώς θα το κάνουμε, πώς θα υλοποιήσουμε κάποια εργαλεία παρέμβασης για να ανταποκριθούμε σε κάποια θέματα. Σε ό,τι αφορά το γάλα τώρα, Νομίζω ότι είπατε ε, κάποια πράγματα, ε, απογοήτευση για αυτό το πακέτο κτλ. Κοιτάξτε, κάποιοι στην Ευρώπη θεωρούν ότι αυτό το πακέτο πάει πολύ μακριά και κάποιοι το αντίθετο. Μα αυτό ακριβώ είναι και το ωραίο στην Ευρώπη. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να πετύχουμε τη συνένεση, το συμβιβασμό. Ιδίω όταν υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετε ε, απόψεις. Αυτό είναι ε, το ενδιαφέρον στην πολιτική, ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειε ε, προσέγγισης, σύγκλησης των διαφορετικών απόψεων. Τώρα, εάν με βάζετε εμένα σαν μεγάλο κορίτσι να γράψω την έκθεση, δεν θα τα έλεγα έτσι βέβαια, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα και να υπάρξει και μια αξιολόγηση. Καλό είναι να λαμβάνονται μέτρα, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθεί και η συνάφειά τους και η αποτελεσματικότητά τους. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν ξέρω ποιος μου έθεσε το ερώτημα συγκεκριμένα για το ποια είναι η θέση τελικά, η οριστική, τελική θέση. Ίσως να μην σας ε, είπα ξεκάθαρα τι έγινε. Δεν θελήσαμε να συζητήσουμε. Επειδή είπαμε ότι δεν είναι βάση συζήτησης αυτό, δεν συζητήσαμε καν. Ετέθησαν κάποια ζητήματα, τα προβλήματα που έχουμε στην κοινωτική αγορά κτλ. Δείξαμε κάποια προβλήματα νομική φύσεω. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει εξέλιξη στο θέμα των ε, γενετικό τροποποιημένων οργανισμών, αλλά δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Όλοι θέλουν το δικό τους. Κάθε χώρα θέλει τα δικά της. Άρα πρέπει μεταξύ των δύο θέσεων να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν το συζητήσαμε το θέμα, δεν τοποθετηθήκαμε να επιταχύνω, γιατί πάει πολύ γρήγορα η ώρα, περνάει η ώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εισαγωγέ προϊόντων. Συμφωνούμε νομίζω, στο ίδιο μήκο κύματο βρισκόμαστε. Φυσικά και τα εισαγόμενα πρώτα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνει ε, μέσω των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Καλό είναι να πούμε και να αναγνωρίσουμε ότι εμείς κοιτάξτε έχουμε πρότυπα που ίσως κάποιες φορές υπερβαίνουν τα πρότυπα αποκλειστικά ασφάλεια των τροφίμων ε, θέλουμε να εφαρμοστούν τα πρότυπα αυτά και στα εισαγόμενα προϊόντα. Ίσως αυτή είναι μια πιθανή οδός. Τώρα, ετικετοθεσία, ποιότητα για τους καταναλωτές, είναι στο πακέτο ποιότητα. Αυτό το σήμα ποιότητας. Νομίζω έχετε εργαστεί και για την ε, ετικετοθεσία της ονομασίας προέλευσης. Τώρα για όλα τα προϊόντα δεν ξέρω αν είμαι 100% υπέρ να υπάρχει αυτή η ετικέτα ε, και ιδίω αν είναι ένας ε, καθαρός εξαγωγές-εισαγωγές δεν είναι εύκολο. Τώρα για συγκεκριμένα Πρώτα ταφική προέλευση, ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά αν θέλουμε να διαβάζουν οι καταναλωτέ και να καταλαβαίνουν τι γράφει η ετικέτα, πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Εάν θέλουμε τεράστιες ετικέτες, ε, ολόκληρα ε, εκατοστά, δεν θα τα διαβάσει όλα αυτά που γράφουν ο καταναλωτής και δεν θα πάρει τις πληροφορίες που πρέπει να πάρει. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη εάν μακρηγόρησα. Καθόλου Σαμπίν, καθόλου, ίσα ίσα. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Πρώτος ε, ε, γεγραμμένος Εύανς Γκαρσία και μετά Ταραμπέλα. Ιεράν Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ε, απελθούσα προεδρεύουσα του Συμβουλίου Γεωργίας. Να την ευχαριστήσω. Ε, πράγματι γίνεται ο απολογισμό ε, του εξαμήνου τη Προεδρία σα και νομίζω ότι το σημαντικότερο που πρέπει να μα απασχολήσει τώρα είναι το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική. Αναφερθήκατε στην έννοια του ενεργού αγρότη. Είναι ενδιαφέρον ο όρο αυτό, αλλά θα είναι ενδιαφέρον και στο βαθμό που αυτό ο ορισμό ε, θα αντιστοιχεί με το στόχο μα. Γιατί ο στόχο μα, τουλάχιστον ο δικό μου στόχο, είναι τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν σε αυτού που είναι πραγματικά αγρότε και που πραγματικά συντηρούν ε, την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Κανένας ε, Νομίζω από τους ε, αγρότες ε, σήμερα ε, δεν έχει επαρκές εισόδημα, δεν δεν, του, δεν έχει τα χρήματα που χρειάζονται. Δεν πρέπει όμως να έχουμε οικονομική εξάρτηση, αλλά ούτε και εξάρτηση από τρόφιμα. Θέλουμε να μπορούμε να περνάμε από τη μια γενιά στην άλλη, θα πρέπει να μπορούμε και να εξασφαλίζουμε την επάρκεια στα τρόφιμα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι να πετύχουμε την ανταγωνιστικότητα. Και για να πετύχουμε την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, δεν πρέπει η παραγωγή μας να, είναι, να πέσουν στη δεύτερη κατηγορία, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο. Γιατί το λέω, ε, γιατί το λέω αυτό, γιατί οι παραγωγοί μας ε, ε, έχουν τόσα προβλήματα, τόσα μειονεκτήματα, τόσες απαιτήσει που πρέπει να, να ικανοποιήσουν, που στον ανταγωνισμό με τρίτες χώρες δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι αδύνατος ο ανταγωνιστός, γιατί πρέπει να πληρώσουν πιο ψηλού μισθούς, τα φυτογενομικά προϊόντα είναι λιγότερα και πιο ακριβά, πρέπει να πληρώνουν πιο, πολύ πιο ακριβά το νερό από τις τρίτες χώρες και γιατί όλες και κάθε μία ξεχωριστά κοινοτικές παραγωγές είναι πιο ακριβές λόγω των απαιτήσεων που εμείς επιβάλλουμε. Αν λοιπόν δεν υπάρξει ισοδυναμία, εξίσωση δεν θα έχουμε κανένα, ε, καμιά άλλη εξέλιξη. Και πώς θα τα εξώσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαιτούμε το ίδιο από τις τρίτες χώρες. Το ίδιο που απαιτούμε δηλαδή από του εθνικούς παραγωγούς. Και αυτοί η απέτηση θα πρέπει να είναι πραγματική και θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό σύστημα ελέγχων. Και θα πρέπει να υπάρχει και πραγματικά να επιτυγχάνει το στόχο του. Από το Συμβούλιο τώρα εγκρίθηκε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο. Εγώ λυπούμαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη σε σχέση με μια έκθεση μάλιστα του Όλαφ που καταδικάζει και καταγγέλει ε, την ε, συστηματική παραβίαση των τιμών εισόδου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχουμε τα επίσημα έγγραφα της Όλαφ που τα έχει η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι πριν μιλήσουμε για το μέλλον θα έπρεπε πρώτα να έχουμε λύσει τα προηγούμενα προβλήματα. Και να πω και κάτι άλλο, το Κοινοβούλιο μας δεν κατάφερε να επιλύσει ένα αίτημα για κάποιες εδαφικές ε, ε, διεκδικήσει κάποια δαφικά θέματα σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας που προβλέπει ε, μείωση κάποιων τιμών για προϊόντα και για, για παραγωγές, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνισή τους. Είναι πολύ άσχημο για τον Νότο, για τη γεωργία του Νότου και είναι πολύ κακό το οποίο ε, εγκρίθηκε και δυστυχώς είναι το κομμάτι της Βελικής Προεδρίας που με λυπεί. Ο κύριος Ταραμπέλα. Και εγώ θα πω το, το, δικό μου ε, καλό λόγο σε αυτό το στεφάνι των κομπλιμέντων που σου έχει απευθυνθεί Σαμπίν. κάνατε πολύ καλή δουλειά ε, απ' την άλλη πλευρά βεβαίως ε, είναι σαφές ε, ότι για να μπορέσει να εκφραστεί είναι, είναι πολύ περιφερειοποιημένη η γεωργική πολιτική στο Βέλγιο και για να μπορέσει να εκφραστεί η, επίτρο, η, συγγνώμη, η Υπουργό θα πρέπει οι Φλαμανδοί και οι Γουαλόνοι να συμφωνήσουν πρώτα. Εν πάση περιπτώσει Ας μιλήσουμε λίγο στο μέλλον. Στην ανακοίνωση, για το μέλλον, στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει μεταρρύθμιση της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής που θα είναι πιο ανοιχτή και βεβαίως αυτό συνάδει και με την ε, νέα προσέγγιση γεωργία, οικονομία, κοινωνία. Ε, δεν θέλω να εστιαστώ στο πρώτο ή το δεύτερο πυλώνα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα περιέχει ο καθένας, αλλά να αναφερθώ σε αυτή την επιθυμία ε, μερικών ε, τα περιβαλλοντικά να μεταφερθούν στο δεύτερο πυλώνα με συγχρηματοδότηση, πράγμα που σημαίνει έστω εν μέρη, αλλά πάντως επαναπεριφερειοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πιστεύω, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι θα πρέπει κάτι να μας πείτε γι' αυτό. Αγορά του γάλακτος επίσης. Μπορώ να πω ότι ενδεχομένως το γεγονός ότι δεν ε, ε, δεν παίζουμε τον ρόλο του χωροφύλακα ε, της, του, του διακανονισμού ενδεχομένως ε, είναι κακό. Ε, ε, περιμένουμε να υπάρχει αυτορύθμιση. Εσείς πιστεύετε ότι η κεντρική εξουσία, η πολιτική εξουσία μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στη ρύθμιση των αγορών. Δύο ξύνες τώρα, μεγάλο κεφάλαιο. Πριν από μερικά χρόνια ε, είχαμε το ίδιο πρόβλημα με την εταιρεία Φερκέστα και νομίζω ότι δεν πρέπει να διστάσουμε να αποκαλέσουμε εγκληματική αυτή την ενέργεια. Εγκληματίες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έλεγχοι λοιπόν, ε, οι έλεγχοι ε, γίνονται ε, σεβαστοί, οι κανόνες γίνονται σεβαστοί από την συντριπτική πλειοψηφία. Υπάρχουν όμως μερικοί εγκληματίες που ξεφεύγουν, μερικοί που, εγκληματίες που παρεκκλίνουν και λόγω αυτών των ολίγων θα πρέπει να βαρύνουμε ακόμα περισσότερο τα, τα, τα πρότυπα και τα στάνταρ. Αλλά για να αποφύγουμε αυτό που είναι ήδη βαρύ και πολύ δεσμευτικό, ε, το πιο δεσμευτικό ίσως ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως δεν θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερους ελέγχους ε, σε αυτές τις επικίνδυνες, ας τις ονομάσουμε, επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Herbert Dorfman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Υπουργό. Θα ήθελα εν συντομία να θίξω τρία θέματα. Καταρχήν το γάλα και όσον αφορά τις ιδέες που ανέπτυξε ο Μάρτιν Χόισλινγκ, ο συνάδελφος, πρέπει να συμφωνήσω μαζί του γιατί ένα από τα προβλήματα του πακέτου αυτού είναι ότι μόνο ο τρεις από τις προτάσεις της ομάδος υψηλού επίπεδου έχουν εφαρμοστεί και ιδιαιτέρως μόνο στην ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των γεωργών Λοιπόν με τη βιομηχανία, χωρίς όμως να θίγουν το τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια. Ε, και κατά αυτόν τον τρόπο παραμένουν περισσότερα χρήματα στη βιομηχανία, αλλά δεν φτάνουν στους γεωργούς. Πράγμα που θα έπρεπε να ε, γίνεται, διότι ε, εάν υπάρχουν συνεταιρισμοί, σημαίνει μένα ότι επειδή στους συνεταιρισμούς ο γεωργός είναι και ο αυτοί έχουν περισσότερα χρήματα από ό,τι σε άλλες ε, περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ολόκληρη την ε, αλυσίδα και πώς θα τη ρυθμίσουμε από τον Γεωργό μέχρι ε, την τοποθέτηση του γάλατος στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στον αγοραστή και να διατυπωθεί μία πρόταση προς όφελος όλων. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ε, ε, ενοποιήσουμε και να ρυθμίσουμε την πολιτική της γεωργίας αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει κανείς να συγχαίει τις προστατευόμενες ονομασίες προελεύσεως και τις ονομασίες τόπου παραγωγής οπότε Επίσης ε, αντιλαμβάνομαι ότι έγινε και μία πρόταση για να ε, ε, προστατεύσει κανείς ε, ε, τις ορεινές περιοχές αλλά τελικά απέτυχε η προσπάθεια αυτή και βλέπω ότι δεν περιλαμβάνεται πλέον ε, ο τομέας αυτός στις νέες προτάσεις. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι ρόλο παίζουν οι γεωργοί, πόσο επηρεάζουν την διαχείριση της ονομασίας προελεύσεως και πρέπει να δούμε πώς πώς ε, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να τοποθετηθούν στην αγορά. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ε, γεωργίας ή μάλλον για να διατυπώσω μία πρόταση, αυτό που με εκπλήσει είναι ότι δεν συζητάμε καθόλου σε αυτά τα συμφραζόμενα τους νέους αγρότες. Δηλαδή έχουμε μία πλειοψηφία νέων κάτω των 35 ετών και κάποια στιγμή θα αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον γεωργοί. Πρέπει λοιπόν επιγόντως να προσπαθήσουμε κάτι να κάνουμε ώστε να προσελκύσουμε τους νέους στη γεωργία και αυτά τα οποία έγιναν μέχρι στιγμή στο δεύτερο πυλώνα δεν επαρκούν διότι οι εμπειρίες κατά τα τελευταία χρόνια απέδειξαν ότι δεν υπάρχει βιώσιμη λύση και θα πρέπει να εντάξουμε νέους στη γεωργία για να μπορέσουμε να έχει μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο τελευταίος εγγεγραμμένος είναι ο κύριος Ανιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αναφέρετε τις δύο τρομελές λέξεις κλιματολογικές αλλαγές που με τρομάζουν. Πρέπει να σας πω τι γίνεται με τα ζαχαρότευκλα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή και την καλλιόργησή τους. Μιλάμε για τη Βρετανική ζάχαρη και ε, στο παρελθόν ε, η γεωργία αυτή αποφάσισαν ε, να επεκτείνουν την περίοδο της καλλιεργίας ζαχάριος και έχουν πληγεί χιλιάδες τώρα διότι ο κάνει πάρα πολύ κρύο και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας. Πρέπει λοιπόν κάτι να ε, σταματήσετε. Εάν θέλετε να ε, κάνει περισσότερο κρύο, κάντε ε, ένα συνέδριο, διότι μετά την Κοπενχάγη έκανε κρύο και μετά από το Κανκούν έκανε ακόμη πιο κρύο. Οπότε ίσως του χρόνου θα μπορέσουμε, μια και δεν έχουμε φέτος συνέδριο, να έχουμε πιο θερμό χειμώνα, διότι τα, οι γεωργοί δεν χρειάζονται να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, συζήτηση, να δώσουμε για μια τελευταία φορά τον ε, λόγο στην κυρία Σαμπίν Λαριέλ ε, για τα τελικά της, τα τελικά της σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από την τελευταία παρατήρηση. Όταν μιλάμε για προπαγάνδα για την κλιματική αλλαγή, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, την ιδέα του. Δεν νομίζω όμως ότι είναι προπαγάνδα όταν λέμε ότι η γεωργία είναι το πρώτο θύμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά εν μέρει ευθύνεται ε, ε, για την κλιματική αλλαγή αλλά μπορεί και να συμμετέχει στην επίλυση του προβλήματος. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό όμω. Σήμερα δεν κάνουμε διάσκεψη για το, για το κλίμα και το κλίμα και οι κλιματικέ αλλαγέ δεν είναι η ειδικότητά μου. Εγώ παρακολουθώ τους επιστήμονες ε, και επίσης κυρίω και την άποψη ενός έγκριτου βέλγου επιστήμονα που ασκεί την πραγματογνωμοσύνη για τη ΖΙΕΚΑ Αυτά. Ε, να απαντήσω και στις τρεις άλλες παρατηρήσεις ε, για την ενεργητική γεωργία. Συμφωνώ μαζί σας, ε, κυρία μου, ότι πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα έννοια ε, πολλοί συνάδελφοι και ε, η Γερμανίδα κυρίως ε, συνάδελφος είπε κάτι ενδιαφέρον. Δηλαδή παρά να ή αντί να καθορίσουμε την έννοια της ενεργητικής γεωργίας δεν θα έπρεπε πρώτα να καθορίσουμε αυτό που δεν είναι γεωργία, δραστηριότητα που δεν αποτελεί γεωργία. Ας πούμε Εάν ε, ε, από ένα μεγάλο χτήμα, ε, ένα μεγάλο κομμάτι έχει γίνει η γήπεδο του γκόλφου, προφανώς δεν μπορεί να ενταχθεί στην γεωργία αυτή η δραστηριότητα. Βεβαίω είναι λίγο καρικατούρα αυτό το παράδειγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες ιδέες και κάποιε συγκεκριμένε ε, αρχές έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε και με το Κοινοβούλιο ε, έτσι ώστε να προσεγγίσουν οι απόψεις μας ή να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να το κάνουν η προβληματική των νέων γεωργών. Συμφωνώ απολύτω μαζί σας κυρία μου ότι έτσι είναι. Εάν θέλουμε να καθορίσουμε μια νέα αντίληψη για την ευρωπαϊκή πολιτική θα θέλουμε οπωσδήποτε να είναι πιο σταθερή, δηλαδή να μην αλλάζουμε κάθε δύο-τρία χρόνια τους κανόνε του παιχνιδιού. Εάν ε, ξεκινήσει αυτή η νέα πολιτική για το 2013, τουλάχιστον να φτάσει μέχρι το 2020, και εν πάση περιπτώσει πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτούμε την ε, νέα, αυτή τη μικρή νέα κοινή γεωργική πολιτική ως ε, ε, υπόβαθρο και τον ρόλο που θα πρέπει και μπορούν να παίξουν οι νέοι γεωργοί, γιατί αυτή είναι το μέλλον της γεωργίας. Γιατί εάν σκεφτόμαστε και συζητάμε και συζητάμε και ξανασυζητάμε και τελικά βρεθούμε με μια χούφτα γεωργούς, τότε πραγματικά δεν έχει έννοια όλο αυτό να ακούμε τους νέους γεωργούς, να, να ακούμε, να προσέχουμε τι ζητούν ε, και να συζητούμε μαζί τους. Τώρα, Εάν ε, ε, ξέρω κι εγώ με τα λίγα, τα φτωχά, τις φτωχές μου γνώσεις για το ποδόσφαιρο, εάν θέλουμε από τη δεύτερη κατηγορία να πάει κανείς ε, στην πρώτη, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει κάποια χρήματα, να κάνει το στάδιο, το γήπεδο του, του ποδοσφαίρου καλύτερο, να αγοράσει καλύτερους παίχτες. Επομένως, είναι γεγονός ότι όσο φιλόδοξα και είναι τα προγράμματά μας και τα σχέδιά μας, εάν δεν έχουμε τον αντίστοιχο προπολογισμό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ε, Απ' την άλλη πλευρά, ευτυχώς ή δυστυχώς δεν θα το αποφασίσουμε σήμερα, η Ευρώπη δεν ζει ε, σε πλήρη αυτάρκεια και βεβαίως αυτού του είδους ε, οι συζητήσεις και οι συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ. Τώρα, γιατί, αυτά που είπατε για το Μαρόκο προηγουμένως, αλλά και τόσα συνέβησαν με τις συμφωνίες Μερκοσούρ, με ενισχύει στην άποψή μου ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πολυμερώς και επομένως επί των πολυμερών συμφωνιών και όχι βάσει δημερών πολυμερών συμφωνιών. Ε, γιατί ε, μία στις δύο φορές μέσω αυτών η βάση, η λόγω αυτών των διμερών συμφωνιών ε, οπωσδήποτε θα πληρώσει τελικά η γεωργία. C'est dedans aussi qu'on doit pouvoir faire reconnaître ailleurs nos normes. Mais c'est aussi pour moi. Τέλος, πιστεύω ότι όλα αυτά ακριβώς μας ε, ε, επιβεβαιώνουν τις φιλοδοξίες μας ε, για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και ξέρουμε ότι θα είναι πιο, θα κοστίζει περισσότερο, θα είναι πιο δαπανηρή, πιο ακριβή η δική μας γεωργία. Μα γιατί είναι πολύ απλό, γιατί εμείς θέλουμε να είναι ανταγωνιστική, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να έχει ευαισθησίες κοινωνικές, ευαισθησίες περιβαλλοντικές, ευαισθησίες κλιματικές κλιματικές κτλ. Και ε, από την άλλη πλευρά, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε τα χρήματα για την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, ακριβώς γι' αυτό χρειαζόμαστε τον προπολογισμό της ΚΑΠ έτσι ώστε να, μπορέσουν, ε, να μπορέσει η γεωργική παραγωγή να αντεπεξέλθει σε αυτές ε, τις ιδιαιτερότητες και σε αυτές τις απαιτήσεις. Τώρα, εάν μου πείτε ότι από αύριο ε, χαμηλώνουμε το γενικότερο επίπεδο των απαιτήσεων, τότε αλλάζει και το ζήτημα του προϋπολογισμού. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σωστές οι ιδιαιτερότητες που έχουμε στην ευρωπαϊκή γεωργία. Και επομένως ε, ε, κατανοούμε γιατί πρέπει να υπάρχουν χρήματα εκτός και αν μου πείτε ότι θα αλλάξουμε εντελώς την ίδια τη βάση της διατροφικής αλυσίδας αλλά στο τέλος θα πληρώσει πάλι ο, ο, ο Ευρωπαίος καταναλωτής, ο Ευρωπαίος πολίτης. Κύριε Ταραμπέλα, σχετικά με το δεύτερο πυλώνα ε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος και ισχυρός ε, πρώτος πυλώνας. Το θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης ε, που μας ενδιαφέρει είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μιλάμε μόνο για σεβασμό του περιβάλλοντος, μιλάμε για σεβασμό του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας, της ευζοίας των ζώων, της υγείας των ζώων, μια σειρά αποθετικά πράγματα. Εγώ θα ε, εξακολουθήσω όμως να υποστηρίζω και να υπογραμμίζω τη λέξη κλειδί που είναι απλούστευση. Απλούστευση της κοινή ζωικής πολιτικής. Και αυτό που θα ήθελα επίσης ε, θα είναι η, τα πράγματα να είναι πιο σαφή. Δηλαδή τι ανήκει στον πρώτο πυλώνα, τι ανήκει στο δεύτερο. Εάν πούμε ότι οι βασικές ε, περιβαλλοντικές απαιτήσει ε, αφορούν τον πρώτο πυλώνα, μέσω πολλαπλής συμμόρφωσης, μέσω άλλου συστήματος, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ε, και να πούμε ότι το δεν τα είναι στο δεύτερο πυλώνα. Αυτό θέλω να είναι σαφή τα πράγματα. Ρωτήστε σήμερα πώς τα καταφέρνει ο κάθε γεωργός σε αυτά τα πλοκάμια, τους δεδάλους μάλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής τι να σας πω, είναι σαν να ψάχνει ψήλο στα άχυρα. Ε, επομένως, απλούστευση και ξανά απλούστευση. Πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τον ε, δημόσιο ρόλο στην ε, ρύθμιση, δηλαδή τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι δημόσιες αρχές στην απλούτευση, Κοιτάξτε, η απόφαση για να σταματήσουν οι ποσοστώσεις λήφθη το 2003, δεν επανερχόμαστε, αλλά οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα πρέπει ο δημόσιος τομέας ε, να στηρίζει κατά κάποιο τρόπο ε, κάποια θέματα. Ε, ναι, επομένως να στηρίζει, να διασφαλίζει την διαφάνεια των τιμών, και αυτό όχι μονάχα σε κάθε χώρα μέλο, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφάνεια λοιπόν. Και η διαφάνεια αυτή επιτρέπει και βοηθάει γενικά, αλλά ε, και βοηθάει τους γεωργούς ε, να έχουν κάποιες συμφωνίες για τις ε, τιμές. Και κατά αυτή την προστακή οδηγούνται και οι προσπάθειες της Κομισιόν. Όσον αφορά την, ε, ε, την, ε, τις ετικέτες. Textuellement ou encadré de façon formelle que c'est exclu. Faudra utiliser une autre voie, mais... ε, τώρα, ναι, μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτούς που σε αυτούς που παράγουν και ειδικά προϊόντα, είτε σε ορεινές περιοχές, είτε ε, ο, οτιδήποτε άλλο ειδικό προϊόν. Ναι, βεβαίως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Ε, τώρα, και για την ε, διοξίνη έχεις δίκιο ότι και η Γερμανία ε, ε, εμείς μάλλον στο Βέλγιο έχουμε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα δηλαδή εμείς υποχρεώνουμε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί ζωικό λίπος να κάνει εκ των προτέρων ελέγχους ε, και βεβαίω ε, εμείς έχουμε ήδη τους ελέγχους αυτούς. Φαντάζομαι ότι και η Γερμανία θα αρχίσει να εφαρμόζει αυτούς τους ε, ελέγχους και βαρύνεται ενδεχομένως η ανταγωνιστικότητά μας, αλλά παρόλα αυτά έτσι πρέπει να γίνει. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Σαμπίν, σε ευχαριστούμε και για όσα μας είπες και για την εργασία της Βελγικής Προεδρίας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ζωηρό τρόπο με τον οποίο μας περιέγραψες τις εξελίξεις στην Γεωργία. Θα ήθελα να καλωσορίσω ένα, μια νέα συνάδελφο, την κυρία Λεγκρούνη, η οποία έγινε πλέον μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Δέκα λεπτά διάλειμμα αναμένοντας τον ε, προεδρεύοντα ε, Σάντορ Φαδέκας. Δέκα λεπτά διάλειμμα.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 Ξαναρχίζουμε τις εργασίες ε, της ε, Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα και εξ ονόματος όλης της Επιτροπής ε, Γεωργίας θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ούγγρο Υπουργό κύριο Ζάντορ Φαζέκας προεδρεύοντα στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2011 υπεύθυνο για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Αγαπητέ Πρόεδρε, υπό την ε, δική σας ε, ε, ηγεσία θα ασχοληθούμε με μια σειρά γεωργικών προβλημάτων. Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, το ζήτημα του γάλακτος και βεβαίως με μεγάλη προσοχή θα περιμένουμε να ακούσουμε την άποψή σας. Επίσης, θα θέλαμε επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την ε, στρατηγική σας ε, σχετικά με την ε, παροχή διατροφικής βοήθειας στους αυτόχθονες. Μας είπαν ότι ακριβώς ένα από τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν μπορέσατε να το συζητήσετε μέχρι τώρα. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, αγαπητέ Σάντορ, για να μας μιλήσετε για την ε, γεωργία στην Ευρώπη. Köszönöm szépen, tisztelt κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μεγάλη τιμή που μπορώ να σας απευθύνω το λόγο σήμερα και να σας ε, μιλήσω για τα θέματα τα οποία απασχολούν την Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μου, αλλά προτού ε, αναφερθώ σε γεωργικά θέματα θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να σας ε, δεχτώ προσωπικά όταν είχατε έρθει το 2010 στη χώρα μας διότι υπήρχε μία πλημμύρα η οποία μας είχε πλήξει και γι' αυτό το λόγο ε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να σας συναντήσω προσωπικά. Σύμφωνα με την άποψη της Ουγγρικής Προεδρίας η Γεωργία συνεχίζει και παραμένει ένα βασικά ευρωπαϊκό θέμα το οποίο ε, έχει συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή να εξασφαλίσει διατροφή εις ε, τους κατοίκους και να προωθήσει και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Για να γίνει αυτό πρέπει να ανταποκριθεί στις διεθνές ε, προκλήσεις, την βιοπικιλότητα, τις κλιματολογικές αλλαγές, τη δημιουργία θέσεων ε, Είμαι είμαι βέβαιος ότι χωρίς μία σωστή γεωργική πολιτική δεν θα μπορέσει να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι μιλάμε για έναν στρατηγικό τομέα ο οποίος είναι πολύ βασικός για όλους μας η γεωργία είναι η πρώτη πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως. Ήδη προ δεκαετιών η γεωργία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για το εσωτερικό της Ευρώπης αλλά και για την κοινή γνώμη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς τη στιγμή όπου ε, πρέπει να σκεφτούμε τη χρηματοδότηση της νέας γεωργικής πολιτικής να έχουμε ένα ασφαλές πλαίσιο χρηματοδότησης. Και επ' αυτόν θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα για τη σημασία της γεωργίας. Η γεωργία απασχολεί ακόμη και σήμερα περισσότερους εργαζομένους από ότι η αυτοκινητοβιομηχανία. Και η Γεωργία ε, καλύπτει ολόκληρο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι βασικό η νέα πολιτική να τελεσφορήσει και η νέα μας εργασία να στεφθεί από επιτυχία. Για να γίνουν αυτά πρέπει ε, και εμείς να κάνουμε ε, προσπάθειες και κατά τη γνώμη μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας βασικός σύμμαχος των κρατών που ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της γεωργικής πολιτικής. Η Ουγγαρία θέλει να έχει μία προεδρία φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σέβεται. Σέβεται τη γνώμη κάθε ε, Επιτροπής. Θεωρεί ότι εσείς είστε οι ομόλογοί μας ε, και πρέπει να συζητάμε από κοινού τα διάφορα θέματα. Τα θεσμικά μας όργανα ε, θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για το επόμενο εξάμεινο και πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα είναι πιο ρεαλιστική και πιο ουσιαστική από ό,τι διαπιστώσαμε τους τελευταίους μήνες διότι το κράτος μου για πρώτη φορά αναλαμβάνει αυτό το βασικό καθήκον και είμαστε υπερήφανοι οι Ούγγροι που αναλάβαμε αυτό το έργο διότι η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και η Ευρώπη είναι κάτι που έχουμε ε, το οποίο αγαπάμε πολύ και γι' αυτό προσλέπουμε στη συνεργασία η οποία όπως σας είπα είναι βασική για την Ευρώπη. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Στην Επιτροπή σας και στο Συμβούλιο ε, γίνονται σοβαρές συζητήσεις ε, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι ε, το περιεχόμενο που υπάρχει στην ανακοίνωση αποτελεί μια καλή βάση για τις ε, κοινέ μας απόψεις και για τη συζήτηση όσον αφορά το μέλλον της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής. Έχουμε διαγράψει ουσιαστικά τρία θέματα. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών του Δεκεμβρίου καταρχήν μιλήσαμε για την αηφόρο παραγωγή τροφίμων. Εχθές έγινε και μία άλλη σοβαρή συζήτηση για την ε, ε, οικονομία με βιώσιμα φυσικά προϊόντα. Επίσης ε, συζητήσαμε μία ισοσκελισμένη εδαφική ανάπτυξη. Δηλαδή βλέπετε ότι εδώ δεν σας ανακοινώνω ήδη αποτελέσματα συζητήσεων διότι πολλά θέματα εκκρεμούν ακόμη και είμαι βέβαιος ότι και στο Συμβούλιο όπως άλλωστε και στην Επιτροπή σας. Η συζήτηση θα καλέψει όλο το πολιτικό φάσμα και θα ενδιαφέρει τους πάντες. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι με την καθοδήγηση του έμπειρου εισηγητή Albert Dess ε, και το Συμβούλιο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις οι οποίες θα προκληθούν από την εισήγηση αυτή και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας στείλει και μία απάντηση στην ανακοίνωση και η εργασία του κυρίου Ντες είναι μία διασφάλιση για την ύπαρξη και τη δημιουργία ενός λογικού ψηφίσματος. Η Ουγγαρία ε, και η κυβέρνησή μου θα προσπαθήσει να ε, εκπληρώσει το έργο της και να οδηγήσει σε συμπεράσματα. Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε ε, να παρουσιάσουμε τον Μάρτιο αποτελέσματα και συμπεράσματα τα οποία θα ψηφιστούν και θα γίνουν αποδεκτά. Και τώρα έρχομαι στα επιμέρους θέματα και ξεκινώ από το γάλα που είναι πολύ σημαντικό για το πρόγραμμά μας και απασχολεί όλη την ευρωπαϊκή δημόσια γνώμη. Θυμόμαστε τη σοβαρή κρίση την οποία αντιμετωπίσαμε το 2009 στον τομέα της γαλακτοκομίας και η παραγωγοί είχαν πληγεί από αυτή την κατάσταση ε, και νομίζω ότι κανένας παραγωγός δεν έμεινε ε, αμέτωχος, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως αντέδρασε και έλαβε μέτρα. Πέραν αυτού, μία ομάδα υψηλού επίπεδου ερεύνησε με τι μέσα και με τι μέτρα θα μπορούσε να επέμβει ε, μακροπρόθεσμα στο μέλλον διότι το ισχύον πρόγραμμα εκπνέει το 2015. Η ομάδα αυτή υπέβαλε τα πορίσματά της πέρυσι τον Ιούνιο και βάσει αυτών των προτάσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτάσεις της. Τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει αναφέρονται σε τέσσερις τομείς ε, ιδίως. Καταρχήν, είπαμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των παραγωγών και ε, της βιομηχανίας επεξεργασίας πρέπει να ενισχυθούν. Ε, τρίτον, ε, θα πρέπει να προωθήσει κανείς τους συνασπισμούς και τέταρτον θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια διότι είναι διαπιστωμένο ότι ε, διαπιστώνουμε από το τέλος του περασμένου έτους μία εξυγίανση του τομέα της γαλακτοτομίας. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα, ούτε ότι έχουν εξαλειφθεί οι αιτίες της κρίσεως, αλλά ε, σημαίνει ότι ε, μπορεί να προστατευτεί η αγορά του γαλακτοτομίας και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να υπολογίσουμε ένα σταθερό πλαίσιο για την ε, ε, γαλακτοκομία για να μπορέσει να προχωρήσει και γρήγορα η σχετική μας πρόταση. Γι' αυτό και ελπίζω ότι με την Επιτροπή σας θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά και ε, προς όφελος ε, εξευρέσεως μιας γρήγορης λύσης και ελπίζουμε ότι αυτό ε, θα μπορέσει να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας με μια υπερψήφιση στην πρώτη ανάγνωση. Ε, όσον αφορά την κτηνοτροφία ε, και την ε, χειροτροφία. Ελπίζουμε ότι και εκεί θα έχουμε αποτελέσματα και πρόοδους, διότι εχθές στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συζητήσαμε ήδη για το θέμα αυτό και ήδη έγινε μία πρώτη συζήτηση. Είμαστε επιφυλακτικοί αλλά είμαστε βέβαιοι ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις της, διότι πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα είναι κοινό και πρέπει να βρούμε την απάντηση από κοινού. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα οριζοντίου αγοράς δηλαδή στις μεγάλες διακοιμάνσεις των τιμών στην ε, γεωργία τις οποίες θα θέλαμε να μετριάσουμε δηλαδή οι εχμές των τιμών και οι ε, ισχυρές ε, διακοιμάνσεις είναι εις βάρος των γεωργών διότι έτσι οι γεωργοί δεν έχουν καμία πρόσβαση σε επιστώσεις. Χρειαζόμαστε μία συντονισμένη αντιμετώπιση των διακοιμάσεων των τιμών και αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε δεν ε, θα μπορέσει να ε, προχωρήσει η παραγωγή, μπορεί να καταστραφεί και έτσι ε, θα κινδυνεύει και η διατροφική ασφάλεια. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να ακολουθήσουμε την ε, πρωτοβουλία του Προέδρου του G20 της Γαλλίας ε, το οποίο συζήτησε το θέμα αυτό εις τα πλαίσια του G20. Και εδώ αναφέρομαι στην ποιότητα των τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό ε, να ε, ε, διατυπώσουμε μία πολιτική η οποία θα επιτρέψει στη γεωργία της Ευρωπαϊκής ενώσεως να αντισταθεί ή στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει κατά τρόπον ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παράγει ποιοτικά προϊόντα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει δύο νομοσχέδια αφενός ε, αναφέρομαι ε, το σχέδιο μία οδηγίας για την πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και δεύτερον για μία ανανέωση ε, των κανόνων εμπορίας των γεωργικών προϊόντων διότι οι γεωργοί βρίσκονται σε μία ασαφή θέση και υπάρχει πίεση. Γι' αυτό και η Προεδρία θα προσπαθήσει να επιτύχει μία γρήγορη πρόοδο στο πακέτο της διατροφικής ασφάλειας. Ελπίζουμε ότι και εδώ θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά προς όφελος ε, της απλοποίησεως και αναγνωρίζοντας τα πρόσφατα γεγονότα διαπιστώσαμε ότι η τωρινή νομική θέση σχετικά με τις ασθένειες θα πρέπει να εξεταστεί διότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας συνομοθέτης και θα πρέπει ε, να να ε, ε, ε, συνεργαστούμε. Ένα άλλο θέμα, οι μέλισσες είναι πολύ σημαντικές για τη γονιμοποίηση και βλέπουμε ότι τελευταίως οι μέλισσες βρίσκονται σε κίνδυνο στην Ευρώπη και προσφάτως έχει υπάρξει μία πρόταση και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του θέματος η οποία παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο εχθές. Θα θέλαμε λοιπόν ε, να οργανώσουμε ε, ένα συνέδριο επί του θέματος αυτού για να μπορέσουν να γίνουν ε, αποδεκτές, αποδεκτά και τα συμπεράσματα του συμβολέου. Άλλο θέμα τώρα ε, πόσο θα μπορέσει να προσαρμοστεί η γεωργική νομοθεσία στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχέδια ε, για κανονισμούς που έχουν υποβληθεί ήδη από πέρυσι και εδώ αναφερόμαστε στις άμεσες πληρωμές ιδίω όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αντιλαμβανόμαστε ότι επί του θέμα θέματος έχουν διατυπωθεί και άλλες προτάσεις για την χρηματοδότηση της κοινή Γεωργικής επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι κύριε Πρόεδρε ότι είσαστε ο εισηγητής για το θέμα αυτό και αυτά τα βήματα θα προλιάνουν το έδαφος για περαιτέρω επεμβάσεις και στους επόμενους μήνες ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία που θα αποτελέσει ένα πρότυπο και για την μελλοντική μας συνεργασία. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ τελικά να μπορέσω να καταλήξω σε ορισμένες γενικές ε, παρατηρήσεις. Καταρχήν χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, θα διευρύνει την τακτική νομοθεσία και στον τομέα της γεωργίας. Δηλαδή εσείς έχετε εμπειρία στο πώς μπορεί κανείς να συνεργαστεί στον τομέα αυτών. Όσον αφορά τη συναπόφαση βλέπουμε ότι τώρα συζητούμε πολύ περισσότερα έγγραφα και αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Προσωπικά εκτιμώ την, τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο πάντοτε έχει αποδειχθεί πολύ θαραλέο και σοφό στα θέματα της γεωργίας. Οι επαφές λοιπόν μεταξύ των οργανώσεών μας έχουν συσφιχθεί κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μία τακτική νομοθετική διαδικασία με αυστηρές προθεσμίες και θα πρέπει να συντονίσουμε τα προγράμματά μας. Κυρίες και κύριοι, εν ολίγης, αυτή, αυτά ήταν τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ουγγρική Προεδρία. Βεβαίως ε, υπάρχουν και πολύ περισσότερες λεπτομέρειες που δεν μπορώ να παρουσιάσω σε μία τόσο σύντομη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και είμαι στη διεύθυνσή σας αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις ή σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πληρέστατη παρουσίαση. Έχω ένα μεγάλο αριθμό βουλευτών που ζήτησαν να, να λάβουν το λόγο. Γι' αυτό θα ζητήσω από όλους να συνεργαστούμε για να οργανώσουμε το χρόνο αγόρευσης. Ξεκινάμε με τους συντονιστές των ομάδων, με πρώτο τον κύριο Ταραμπέλα. Για άλλο θέμα θέλετε το λόγο. Α, μάλιστα. Επομένως, Άλμπερτ Ντες, πρώτος ομιλητής, πρώτος συντονιστής. Ε, ε, ευχαριστώ Πάολο. Ε, σε, σε Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ, σας συγχαίρω για την ανάληψη της Προεδρίας και όπως είπατε και εσείς ελπίζω ότι κατά το εξάμεινο αυτό θα συνεργαστούμε καλά διότι είχα έρθει και εγώ στην Ουγγαρία και διαπίστωσα την, και ενημερώθηκα για την κατάσταση της γεωργίας στη χώρα σας και μπορώ να επαναλάβω αυτό το οποίο έχει λεχθεί πολλές φορές τελευταίως ότι ορισμένα αυτά τα, από αυτά τα θέματα θα εσωματωθούν στην επόμενη εισήγηση διότι βλέπω ότι στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχουν πολύ διαφοροποιημένες καταστάσεις και ε, έχω προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσα να συγγράψω ένα τεράστιο τόμο. Πρέπει όμως εδώ σαν ε, ευρώ πει πολιτική να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη και την Ευρώπη στο σύνολό της αλλά και ε, θα σέβεται τις ιδιομορφίες του κάθε κράτους. Γι' αυτό και σας είμαι ε, ευγνώμων όπως είπε άλλωστε ε, και η Βέλγιδα υπουργό ότι θα διατηρηθεί το σύστημα των δύο πυλώνων και ότι όλα αυτά θα ρυθμιστούν με τον απλούστερο δυνατόν τρόπο διότι στις επόμενες μέρες θα δούμε πόσο θα διαμορφωθεί η έκθεση κατά τρόπον ώστε να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαμορφωθεί η κοινή γεωργική πολιτική κατά τρόπον ώστε να καταλήξουμε σε μία σαφή νομοθεσία πρόταση για τη γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να παραμείνει η όλη διαδικασία διάφανη διότι διαφορετικά ε, θα πρέπει ε, να ε, παραβλέψουμε την εργασία μας που θα είναι κρίμας. Ίσως κάποιος παράγει τρόφιμα αλλά και ενέργεια και πρέπει να ε, υπάρχει μία βιώσιμη καλλιέργεια όλων των ε, ευρωπαϊκών εδαφών και εγώ τουλάχιστον θα φροντίσω να υπάρξει έξυπνη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, από την ομιλία σας επιτρέψτε μου να σας επισημάνω διάφορα θέματα που δεν, υπήρξε μία σαφής απάντηση και δεν είχε διευκρινίσει και ο Επίτροπος Τσόλος. Μιλάμε για τους μικρούς γεωργούς στην Ευρώπη και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν μικροί γεωργοί στην Ελλάδα με ε, μερικά ε, σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ή στην ε, Λετωνία υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός εκταρίων και θα πρέπει πέντε της 100 των πόρων του πρώτου πυλώνα να αποδοθεί στα κράτη-μέλη επιπροσθέτως για να μπορέσει κάθε κράτος μέλος να προβεί στο δικό του ορισμό των μικρών γεωργών και να μην παραμείνει αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης μιλάμε και για τα ανώτατα όρια στην Ευρώπη και έχω διαπιστώσει ότι και εδώ πρέπει να καθορίσουμε ακριβώς ποιο θα είναι το ανώτατο επίπεδο και ίσως θα έπρεπε να γίνει μία πρόταση από εσά και να αξιολογήσετε σαν Ούγκρος πώς βλέπετε το θέμα. Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών, νομίζω ότι από τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη αντελήφθην ότι τα κράτη θα θέλουν να υπάρχει μία κελισμένη πολιτική αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι ε, κάθε κράτος θα πρέπει να υπολογίσει τι συμψηφίζεται μεταξύ πρώτου και δευτέρου πυλώνα και μετά ε, να κατολίξουμε σε ένα συμπέρασμα για να έχουμε μία υγιή βάση υπολογισμού. Πέραν αυτού θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχουν μόνο διαφορές για τις αντισταθμιστικές ε, ε, ε, πληρωμές αναπηλώνα μεταξύ κρατών μελών αλλά και εντός ενός κράτους μέλους. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στο ίδιο κράτος διαφορές μεταξύ αντισταθμιστικών πληρωμών από 5 έως 50 ευρώ. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη δικαιοσύνη και στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και θα προσπαθήσουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατυπώσουμε τις σωστές απαντήσεις. Χαιρετίζω ιδιαιτέρως ότι είπατε ότι προσβλέπετε σε μια καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αυτή την Επιτροπή και στους επόμενους ε, μήνες θα συνεργαστούμε και έτσι εγώ εύχομαι προς ε, όφελός μας στην Ουγγρική Παροεδρία καλή επιτυχία. Λουίς Κάπουλα Σαντόσα, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω βεβαίως χαιρετίζοντας τον κύριο Υπουργό και ευχόμενος ευόδοση των εργασιών του και μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να θέσω συγκεκριμένα ερωτήματα. Συνήθως ε, σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την παρουσίασή σας, αλλά να μιλήσουμε επί συγκεκριμένου. Πρώτα απ' όλα, με ποιο τρόπο συγκεκριμένο και αυτό βλέπετε και αναγυγνώσκετε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας στα θέματα που μας ε, αφορούν. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, θα έρχεστε κάθε, ενώπιόν μας ε, ε, κάθε φορά που θα έχει Συμβούλιο Υπουργών πριν μετά για να κατανοήσουμε καλύτερα τα πράγματα. Είστε έτοιμος επίσης ε, να δεχτείτε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο. Έστω και αν υπάρχει ήδη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων έχουν παραμείνει σε άτυπο επίπεδο. Με ποιο τρόπο δηλαδή προτίθεστε να εμπλέξετε ε, το Κοινοβούλιο άμεσα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ε, μια πραγματική, σωστή και πλήρη συνεργασία. Και άλλη συγκεκριμένη ερώτηση να σας θέσω. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά ε, την συγκυρία. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί έρχεστε από μια χώρα η οποία οποία παράγει πολύ χείριο κρέας και ξέρετε ότι ο τομέας της ε, χειροτροφίας ε, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία θα πρέπει σύντομα να ανατρέψουμε αν θέλουμε πραγματικά να ανασχετήσουμε, να ανασχετήσουμε, συγγνώμη, να ανασχέσουμε την ε, κρίση. Τι μέτρα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε. Όσον αφορά την τιμή των σιτηρών, το είπατε ότι πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τις υπερβολικές διακυμάνσεις σε τιμών. Ποιες προτάσεις κάνετε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής ε, Πολύ σημαντικό ζήτημα και επ' αυτού έχω συγκεκριμένα ερωτήματα να θέσω. Πρώτον, δίκαιη κατανομή των, ε, της βοήθειας. Συμφωνώ με τον Υπουργό ότι πρέπει να παρακολουθούμε λίγο την κατάσταση και τη συμφωνία Γερμανίας-Γαλλίας. Αλλά υπάρχει και ένα ουσιώδες ζήτημα. Δηλαδή η διατήρηση του status quo όσον αφορά ε, τα, το, το χρηματικό, το οικονομικό ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα η καλύτερη, πιο ισοδίκαιης κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, συμφωνείτε ναι ή όχι ότι το κριτήριο της απασχόλησης και των θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πέρα από το καθαρά περιβαλλοντικό ε, ζήτημα. Βεβαίως ε, πρέπει να άμεσα ή και έμεσα να στηρίξουμε τις θέσεις απασχόλησης. Αυτά ήθελα να πω. Πολλές ερωτήσεις ήθελα να θέσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της ε, Ουγγρική Προεδρία που ήλθε στην Επιτροπή μα και μας ε, εξέθεσε ξεκάθαρα τις προτεραιότητες της και βλέπω και εγώ στη στενή συνεργασία που θα έχουμε το επόμενο εξάμεινο. Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα σημεία κυρίως σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ποια είναι η αποψή σας σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί προϋπολογισμού που θα έχει μεγάλη σημασία και ίσως και επηρεάσει και την ίδια την έκβαση της ε, μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Και υπάρχει και πρόθεση να παγώσει ο προπολογισμό ε, το 12 έως το 2020. Εστάλει μια επιστολή στον ε, Μπαρόσο σχετικά. Τι άποψη έχετε εσείς, ποια είναι η άποψη της Προεδρίας. Δεύτερο ερώτημα διότι υπάρχει πίεση και για περικοπές στον προπολογισμό, αλλά και για περιστολή των πολιτικών της κοινής γεωργικής πολιτικής σε σχέση με τον προπολογισμό. Σίγουρα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις αν θέλουμε να υπάρχει ένας δίκαιος επιμερισμός, μια δίκαιη κατανομή. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την δικαιότερη κατανομή των πόρων μεταξύ κρατών μελών, άμεσες πληρωμές ε, για τη γεωργική ανάπτυξη κτλ. Και ένα τελευταίο σημείο. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε τον τρόπο, πώς αντιλαμβάνεστε τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο Γεωργίας. Πώς προχωρούν οι συζητήσεις αυτές, τι στόχους έχετε για την εκπόνηση μιας θέσης, ενός σχεδίου θέσης μέχρι το Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε να υπάρχει ένα έγγραφο που το έχουν υπογράψει όλοι δεν θυμάμαι, δεν ξέρω μάλλον κατά ε, πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση τον Ιούλιο ή το φθινόπωρο. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση από τους υπουργού που θα λένε τις απόψεις και θα με ενδιαφέρει να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Μπορείτε να πετύχετε συμφωνία πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες που έχετε. Μάρτιν Χόσλινγκ, παρόλα. Ο Μάρτιν Χαϊσλινγκ έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, διότι ήρθατε σε μια πολύ αποφασιστική ε, φάση. Έχετε την Προεδρία της Ενώσεως και σωστά αναφέρατε τα θέματα. Είπατε ότι είναι βασικός ομόλογός σας το Κοινοβούλιο, που μπορεί όμως να είναι και αυστηρός κριτής. Ο διάλογος όμως θα πρέπει να συνεχιστεί μεταξύ μας για το επόμενο εξάμεινο και ε, θα πρέπει να δρομολογήσουμε σωστά τις συζητήσεις μας. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς, πώς εσείς πιστεύετε ότι θα παρουσιάσετε το, τη δέσμη των μέτρων που θα λάβετε. Ε, αναφερθήκατε σε θέματα περιβαλλοντολογικά πώς θα διεκπαιρεώσετε και το θέμα των θέσεων εργασίας και αυτό έχει ε, ερωτηθεί θέλετε αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσετε δυναμικά ή πιστεύετε ότι είναι παρελκόμενα τα οποία ενδεχομένως θα συζητηθούν επίσης Είπατε ότι για το γάλα υπάρχει μια εξυγίανση του τομέα, πράγμα όμως το οποίο μπορεί να μεταστραφεί πολύ γρήγορα, διότι πριν από την τελευταία κρίση υπήρξε μια κατάρρευση των τιμών ε, και εάν υπάρξει αύξηση της παραγωγής μπορεί και να, αυτό να ξανασυμβεί. Θεωρείτε ότι τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικά, όπως έχει ε, ζητήσει επανειλημμένως η Επιτροπή μας ιδίω προς όφελος των γεωργών. Επίσης με ενδιαφέρει στο θέμα που θίξατε σχετικά με τις συνενώσεις και ε, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των γεωργών. Ε, έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα τώρα για τη διοξίνη και υπήρξε μια συζήτηση επ' αυτού ε, και μια αμφισβήτηση αν είμαστε στο σωστό δρόμο στη γεωργική πολιτική. Τι τρώνε τα ζώα μας και αυτό επηρεάζει τον καταναλωτή, τουλάχιστον συζητιάται στη Γερμανία. Ε, όσον αφορά την ασφάλεια των ε, ζωοτροφών, συμφωνείτε με πολλούς που πιστεύουν ε, ότι πρέπει να ζούμε ε, και να ταΐζουμε στα ζώα μας στην Ευρώπη ό,τι παράγεται στους αγρούς μας. Ε, πώς αντιμετωπίζεται το έλλειμμα λευκόματος στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση διότι νομίζω ότι είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητήσετε το επόμενο εξάμεινο και ελπίζω να υπάρχει ένας αμοιβαίος διάλογος κατά τρόπον ώστε να στερθεί, με επιτυχία στο τέλος η Ουγγρική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ Λορέντζο Φοντάνα. Και εγώ χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ελπίζουμε ότι στους επόμενους μήνες η συνεργασία μας θα είναι καρποφόρα. Πολλά ερωτήματα ήδη έθεσαν οι συνάδελφοι, αλλά μπορώ να είμαι σύντομος. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της ποιότητας των ε, προϊόντων στην Ευρώπη. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ε, ζητήματα ε, τα οποία προτίθεστε από ό,τι ξέρουμε να προωθήσετε και ε, σχετίζεται και με την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας τι θα κάνετε όσον αφορά τις ετικέτες και επίσης τι θα κάνετε απέναντι στις τρίτες χώρες από τις οποίες εισάγουμε γεωργικά προϊόντα. Γιατί γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι δεν είναι οι ίδιοι οι κανονισμοί που διέπουν τις χώρες αυτές. Εμείς έχουμε πολύ πιο δεσμευτικές αρχές, πολύ πιο δεσμευτικούς κανόνες με αποτέλεσμα να προκύπτει στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, και να προκύπτει επίσης μεγάλη δυσκολία στους δικούς μας γεωργούς σε σχέση με τους παραγωγούς αυτών των χωρών. Ο Αντιπρόεδρος Βασεβόσκη τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση της ουγγρικής προσέγγιση σε σχέση με τα μελλοντικά συστήματα της κοινή γεωργικής πολιτικής με χαρά άκουσα ότι η Ουγγαρία, μια χώρα η οποία προσδίδει μεγάλη σημασία στη Γεωργία, προεδρεύει σε αυτούς τους δύσκολους, αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ε, το Συμβούλιο Γεωργίας. Ε, τρία ερωτήματα. Το πρώτο, το οποίο τέθηκε από άλλους, ε, είναι το πλαφόν στις πληρωμές. και το θέμα των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών Πώ θα εξομαλυνθούν οι διαφορές που είναι σημαντικές, το γνωρίζουμε. Ίσως, δεδομένων ε, των λίγων πόρων, μακάρι να ήταν περισσότεροι, αλλά δύσκολο το βλέπω, τι πιθανότητες υπάρχουν, ε, τι μηχανισμοί υπάρχουν για καλύτερη ε, εξισορρόπηση. Τώρα, δεύτερο, γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί. Η Ουγγαρία τα κατάφερε καλά στη συζήτηση με τον Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προάσπισε τις περιοριστικές της διατάξεις στι επαφές που είχε με την Επιτροπή. Μήπως θα μπορούσε η Ουγγαρία να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες. Και σε ό,τι αφορά την απλούστευση της κοινή γεωρικής πολιτικής, έχουμε την έκθεση Άσφορτ, την οποία εγκρίναμε εδώ στο Κοινοβούλιο για να δούμε πώς μπορούμε να εξορθολογήσουμε, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να την κάνουμε πιο φιλική προς τον αγρότη, την κοινή γεωργική πολιτική. Προβλέπετε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία ως Ουγγρική Προεδρία. Αν δηλαδή δεν αλλάξει το status quo των αγροτών, να μην χρειάζεται να κάνουν τις αιτήσει τους ε, κάθε χρόνο, αλλά να υπάρχει μια πολυετής προσέγγιση και να είναι και λιγότερο περιοριστικές οι ποινές ε, και τα πρόσημα, γιατί είναι περιοριστικό το σύστημα, πολύ περιοριστικό. Και θέλουμε να τονίσουμε ότι κάποιες φορές οι αγρότες ε, τιμωρούνται αχρίαστα, υφίστανται πρόστιμα και κυρώσεις. Τι έχετε να πείτε και γι' αυτά. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο γύρος, μάλλον όχι τώρα θα ολοκληρωθεί ο γύρος των ε, συντονιστών ε, με τον τελευταίο μιλητή. Ευχαριστώ, μπετε Ζήτησα, δεν ζήτησα το λόγο. Grazie. Allora adesso darò la parola al Ministro. Ωραία, θα δώσω λοιπόν ξανά το λόγο στον Υπουργό κύριο Σαντόρ Φαζέκας να απαντήσει στις, ε, ε, στις ερωτήσεις και μετά θα ξαναέχουμε γύρω ο, ε, ο, ερωτήσεων αλλά έχουμε ακόμα 20 εγγεγραμμένους, ε, συγγνώμη 14 εγγεγραμμένους, δεν θα έχουμε το χρόνο. Παρακαλώ πολύ να μην ξεπερνάτε το χρόνο αγόρευσή σας για να προλάβουμε. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ και για τα πολλά ερωτήματα. Δεν είναι εύκολο να απαντήσω σε όλους, οπότε ε, θα πρέπει και να σεβαστώ τον περιορισμένο χρόνο μου και ε, τα ερωτήματα χρειάζονται πιο εκτενείς απαντήσεις. Γενικώ όμως η κοινή γεωργική πολιτική δεν ε, είναι τόσο ελεγχόμενοι ώστε ε, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι διαφέρει το μέγεθος των επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά τους και αυτό το είδαμε στις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης ε, έχουμε ε, άλλα στοιχεία. Το σύστημα των δύο πυλώνων στηρίζεται από τα περισσότερα κράτη και είναι πολύ βασικό εδώ να έχουμε ε, σαφείς στόχους, να τους διαχωρίζουμε και να προωθούμε κάθε θέμα χωριστά. Συμφωνώ ότι η παραγωγή και η γεωργή θα ήθελαν ένα πιο σαφές και διαφανές σύστημα αλλά ε, θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία αλλά υπάρχει όλο και περισσότερη ε, γραφειοκρατική εργασία ε, για να υπάρξει δημοκρατία. Βέβαια θέλουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία και να απλοποιήσουμε το σύστημα σύστημα διότι ο γεωργός σύστημα πρέπει να ενταχθεί σε 10-20 συστήματα ενώ ο υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ειδικό για ένα θέμα μόνο, δηλαδή η γραφειοκρατία είναι μεγάλη για τους γεωργούς και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε επικοδομητική πρόταση προς την Ουγγρική Προεδρία. Όσον αφορά τους μικρούς παραγωγούς και τη στήριξή τους, είναι πρόωρο τώρα να προκαταλάβουμε τις αποφάσεις των συζητήσεων στο Συμβούλιο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει ε, να προωθήσουμε τους μικρούς γεωργούς και μόνο ε, εάν συνενωθούν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Βέβαια όλα αυτά είναι ε, θέμα ορισμού διότι το μέγεθος της επιχειρήσεως ε, εδώ μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος στο άλλο και είναι πολύ βασικό κάθε κράτος μέλος να έχει τη δυνατότητα να προβεί στον δικό του ορισμό έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά η ε, οικονομία όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα και τα κράτη-μέλη έχουν υπάρξει επιφυλακτικά. Η συζήτηση ακόμη δεν έχει καταλήξει επί του θέματος αυτού στο Συμβούλιο, αλλά οι βασικοί ορισμοί πρέπει να διευκρινιστούν. Όταν μιλάμε για χώρο, για απασχόληση, για παραγωγή και θέλουμε να αποφασίσουμε, πρέπει να ε, μπορέουμε να διευκρινίζουμε πώς συνδυάζονται αυτά τα κριτήρια. Διότι πολλές φορές δεν ξέρουμε αν τα υπολοιπόμενα κεφάλαια πρέπει να αποδοθούν στα κράτη-μέλη, να παραμείνουν εις τον κοινοτικό προϋπολογισμό για επόμενη χρήση. Ένας στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι να υπάρξει μία ε, αναβίωση της απασχόλησης ή στην ύπαθρο και το θέμα αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Όσον αφορά την δίκαια κατανομή εντός των κρατών μιλών, μελών πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ε, δεν έχει ακόμη διεξαχθεί. Όσο δεν αναφορά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλάμε για μια πιο δίκαια κατανομή, αλλά δεν έχω ψευδεστήσεις, θα υπάρξει συζήτηση. Ο συνδυασμός με τη συνθήκη της Λισαβόνας και συγκεκριμένα με το ερώτημα του πώς θα μπορέσουμε στο μέλλον να συνεργαστούμε επικοδομητικά, Είμαι βέβαιος ότι με τον πρόεδρο θα παραμείνουμε σε συνεχή επαφή ε, ε, επισήμως αλλά και ατύπως για να προωθήσουμε τη συνεργασία μας. Υπήρξε κι άλλο ένα ερώτημα. Για την ε, κτηνοτροφία και την κρίση του ειρηνού κρέατος και ε, για το δίχτυ ασφαλείας το οποίο πρέπει να προστατεύσει τους παραγωγούς. Είναι μια μακριά συζήτηση η οποία διεξάγεται και εντός των κρατών μελών και μεταξύ παραγωγών. Η Ουγγρική Προεδρία στηρίζει την εισαγωγή του δίχτυ δικτύου ο ασφαλείας κατά τρόπεν ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις ε, των ε, φυσικών καταστροφών και ε, άλλων δεινών. Χρειάζεται λοιπόν ένα τέτοιο αποτρεπτικό μέτρο το οποίο όμως θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ποικιλομορφία των αγορών και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα συμφέροντα των καταναλωτών, των παραγωγών και να εξετάσουμε με το θέμα πολύ προσεκτικά. Όσον αφορά την ομάδα υψηλού επίπεδου του Συμβουλίου θα την εμπλέξουμε σε αυτή τη συζήτηση διότι υπάρχει ε, και άλλη πρόκληση να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ε, πλημμύρες, στις φυσικές καταστροφές που μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο κίνδυνο για ορισμένες περιοχές της Ευρώπης και μπορεί να διακινδυνεύσουν όχι μόνο την διατροφική προμήθεια αλλά και την παραγωγή τροφίμων διεθνώς. Άρα οι μορφές της παραγωγής θα πρέπει να προστατευθούν έναντι των ε, ακραίων ε, διακυμάνσεων ε, για να μπορούν και οι παραγωγοί να επιβιώσουν των δύσκολων περιόδων και να τροφοδοτούν την Ευρώπη και τον κόσμο με υγιή διατροφικά προϊόντα. Ψάχνω τώρα να βρω ποια ήταν η επόμενη ερώτηση. Ήδη ανέφερα ότι η απασχόληση είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα μας απασχολήσει και έτσι προχωρώ στην επόμενη ερώτηση, δηλαδή τη σχέση του ε, συνδυασμού μεταξύ κοινής γεωργικής πολιτικής και προϋπολογισμού. Ε, όντως, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα κλειδί, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορέσει να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Είμαι βέβαιος ότι η γεωργική πολιτική μπορεί μόνο να επιτύχει αν έχει την αναγκαία χρηματοδότηση η οποία θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Άρα είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί των στόχων και επί των μέσων που διαθέτουμε διότι αν καθορίσουμε σαν ένα σύνολο στόχων τη γεωργική πολιτική και εκεί προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ε, μέσω αυτού του στόχου την διατροφή αλλά συγχρόνων την ανάπτυξη της υπέτρου, στην βελτίωση των όρων διαβίωσης του πληθυσμού της υπέθρου και άλλα θέματα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι θα πρέπει να βρεθούν τα αναγκαία ε, δημοσιονομικά μέσα αλλά θα πρέπει να ε, υπάρξουν καινοτόμες ιδέες και αυτό άλλωστε ε, συνδέεται επίσης με τον προϋπολογισμό. Είναι λοιπόν πολύ πολύ σημαντικό ο προϋπολογισμός να μην μειωθεί. Βέβαια δεν θέλω να προκαταλάβω τα πορίσματα μιας συζήτησης, αλλά πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η κοινή γεωργική πολιτική είναι ίσως η παλιότερη κοινή πολιτική της Ευρώπης. Όσον αφορά τώρα την ε, σωστή κατανομή, ε, έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό. Ο κύριος Λάιον ρώτησε επίσης Ποιες είναι οι προοπτικές ε, για το Συμβούλιο Γεωργίας και ποιος είναι ο στόχος που επιζητούμε. Όπως σας είπα, θα θέλαμε τα συμπεράσματα να μπορέσουν να ψηφιστούν το Μάρτιο, στις συνεδρίες του Μαρτίου, διότι ήδη έχει γίνει προεργασία και ορισμένες σημαντικές φάσεις έχουν διεκπαιρεωθεί. Άλλο θέμα, όσον αφορά την ε, ε, κατανομή και την αναθεώρηση του πρώτου πυλώνα. Έργο του κάθε Προεδρού είναι να διαγράψει τις προτεραιότητες. Με ρωτήσατε λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Η γνώμη μας είναι να διοχετεύσουμε την τις διάφορες γνώμες στη σωστή κατεύθυνση και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των απόψεων των διαφόρων χωρών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή διαπραγμάτευση και να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις που να ικανοποιούν όλους και που θα εξασφαλίσουν την ανανέωση της γεωργικής πολιτικής. Έρχομαι τώρα στο θέμα του γάλατος που είναι ένας πολύ βασικός τομέας ως Όσον αφορά το γάλα και τα προϊόντα γαλακτοκομητά έχουν μεγάλο ρόλο σε πολλές χώρες. Είναι δηλαδή ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και οι μεγάλες διακοιμάνσεις των τιμών μπορούν ε, να βλάψουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στις τιμές του γάλατος. Τώρα, το εάν το πρόγραμμα των μέτρων που έχει καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα επαρκέσουν ή όχι, δεν μπορεί να λάβει απάντηση ακόμη. Θα δούμε θα δούμε στο μέλλον. Αλλά η κατάσταση όπως είπα είναι σταθερή. Και το τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Διοξίνες. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Okay. Ε, είναι πολύ σωστό ότι πρέπει να ταΐζουμε τα ζώα μας με υγιείς ζωτροφές και ε, να μην ε, ε, θέτουμε σε κίνδυνο ούτε την υγεία των ζώων ούτε των ανθρώπων που τρώνε το κρέας αυτό. Το σκάνδαλο της διοξίνης δεν το ακούω για πρώτη φορά διότι πήγα στο Βερολίνο και άκουσα το θέμα αυτό επανειλημμένος. Ε, κάποιοι παρέβλεψαν τη νομοθεσία και αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν για παραδειγματισμό αλλά υπάρχει και άλλο ένα μάθημα που αποκομίζουμε για το μέλλον και το μάθημα αυτό είναι το εξής. Το σύστημα της ε, ε, υγείας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά μέχρι τώρα και υπάρχουν ε, οι αναγκαίοι μηχανισμοί για να εμποδίσουν να φτάσει το μολυσμένο κρέας στο τραπέζι του καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι το Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αποφασίσει να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα. Εχθές ο Επίτροπος Ντάλι ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων που θα εξασφαλίζει καλύτερο ε, ε, έλεγχο των ζωοτροφών και το θέμα που συζητήθηκε ε, επίσης εχθές στο Συμβούλιο είναι ότι θα ληφθεί μία απόφαση σχετικά με τις ιδιωτικές αποθήκες ζωοτροφών. Ε, θέλω επίσης να σας πω ότι η αγορά των χοιρινών είναι κάπως χαλαρή και δεν υπάρχουν επαρκή ε, μέσα που να ε, αναφέρονται στην εμπορία αλλά μέχρι στιγμής είχαμε αποτέλεσμα. Έχουμε όμως και πολλές εισαγωγές και βλέπουμε ότι οι κανόνες για τις εισαγωγές και εξαγωγές δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν της κρίσεως και ε, κάθε μερικά χρόνια έχουμε μία υπερπαραγωγή που θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση της αγοράς. Και αυτό οδηγεί σε μία οπισθοδρόμηση του ζωικού κεφαλαίου. Η αγορά ε, κυμαίνεται και ε, η ε, Βελγική Προεδρία ήδη προετοίμασε την εργασία την οποία εμείς συνεχίζουμε και ε, στις 17 Μαρτίου θα υπάρξει η πρώτη συνεδρίαση όπου θα συζητηθεί κατά προτεραιότητα το θέμα αυτό διότι διακυδεύεται η διαφάνεια των θεσμών. και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους, την νομοθεσία σχετικά με τις ζωοτροφές. Ε, όσον αφορά τις ιδιωτικές αποθήκες, η οποία ε, έχει ε, ξεκινήσει αποτελεί ένα ειδικό μέτρο το οποίο θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος. όσον αφορά τις προδιαγραφές ποιότητος των τρίτων χωρών και ακόμη και των ευρωπαϊκών χωρών είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Όλους όσοι ε, παρίστανται στην αίθουσα αυτή. Διότι όλοι έχουν αγοράσει προϊόντα από τρίτες χώρες τα οποία έχουν τύχει περαιτέρω επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν ε, δύο ήδη τροφίμων. Στην Ευρώπη υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος, μεγαλύτερη πιστότητα στην ποιότητα, μεγαλύτερα προβλήματα και δυνατότητα επιλύσεως των προβλημάτων που πρέπει να λυθούν για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει. Αλλά στην αγορά υπάρχουν και άλλα και ε, άλλα μέτρα και δεν ξέρω αν αυτά συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία διότι η νομοθεσία αυτή συνεπάγεται περισσότερο κόστος, περισσότερο χρόνο που χρειάζεται και ε, θα έπρεπε ε, να λάβουμε υπόψη ότι και τρίτες χώρες ζητούν ευρωπαϊκά προϊόντα να σέβονται τις προδιαγραφές και τις νομοθεσίες τους. Άρα είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτό όσον αφορά το πακέτο ποιότητος των τροφίμων που προβλέπονται δύο οδηγίες όσον αφορά τα προϊόντα ποιότητος, ο χαρακτηρισμός, την ε, ε, σήμανση, ε, τα προϊόντα γεωγραφικής προελεύσεως, η αναφορά στα γεωγραφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά τους, τις ΕΠΕ, είναι ένα πολύ λεπτό τομέας και ε, Θέλω εδώ να αναφερθώ και στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, το θέμα αυτό θα πρέπει να ανοίξει προς ε, την ε, δημοσιότητα όσον αφορά δηλαδή την παραγωγή και την εμπορία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και ελπίζω εφόσον επεξεργαζόμαστε το σημείο αυτό ότι θα πετύχουμε. Θα μπορούσα να σας μιλήσω και για άλλα θέματα και σας ενημερώσω αλλά καλύτερα είναι να ε, απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ γιατί υπήρξατε πολύ λεπτομερείς ε, και φαντάζομαι ότι απαντήσατε ενδελεχώς σε πολλές ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω ότι επειδή αναφέρθηκε σε πολλά θέματα ο κύριος Υπουργός, να περιορίσετε λίγο τις ε, ερωτήσεις σας. Ε, Ταμπάζω, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση που μπορείτε να απαντήσετε εύκολα. Πιστεύετε ότι η πολλαπλή συμμόρφωση πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2014 δηλαδή να υπάρχει μεταφορά πόρων από, την, από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο και στηρίζει αυτή την προσπάθεια η Ουγγαρία. Δεύτερον όσον αφορά ε, ε, τις φορές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πώς ε, μπορούμε να τις απαλλάξουμε από την υπερβολική γραφειοκρατία πώς δηλαδή θα μπορέσει κανείς να διευκολύνει τους γεωργούς και να τους υποκινήσει να προστατεύσουν το περιβάλλον, πράγμα το οποίο ε, είναι αντιφατικό ή στον πρώτο πυλώνα όπου δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των γεωργών. Μεταξύ δηλαδή του τι προβλέπετε και τι όντως γίνεται. Μήπως θα έπρεπε αυτό το θέμα να εξεταστεί κάπως διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χέραντς Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι σίγουρα υπάρχουν τομεί που πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα. Ο πρώτο είναι τα πτηνά και δεύτερον, ε, μεταξύ άλλων, ο χείριο τομέα. Σε ό,τι αφορά τα πτηνά, το ερώτημά μου είναι τι πιστεύετε για τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν προσεγγίζει αυτήν του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ε, τους ε, κλωβούς ομπλωτισμένους και δεν λαμβάνει υπόψη την ε, σύσταση ε, του Κοινοβουλίου ώστε να βοηθήσει εκείνες επιχειρήσεις που προβαίνουν ε, σε αναπροσαρμογή των κλοβών. Τώρα για το χείριο κρέας δεν θα ήταν καλό να πούμε ότι οι ζωοτροφές με ζωικό λίπος όπως από το 2007 σε έκθεση της Επιτροπής για την Ασφάλεια των Τροφίμων τι ε, πιστεύετε λοιπόν αν αυτά ε, τα λύπη θα μπορούσαμε να τα απαγορεύσουμε για, τα για το χείριο κρέας. Είναι άμεση ερώτηση. Ο κύριο Μάτο και μετά κύριε Μαγκίνας. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι θα πρέπει να είναι ένας εταίρος προτεραιότητας στο Κοινοβούλιο θα ήταν καλό και εσείς να είστε εταίρος πολύτιμος για το Κοινοβούλιο και να είστε και ένας ευεργέτης ε, των γεωργικών ε, περιοχών. Τρία θέματα είναι σημαντικά κατ' εμέ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να δεσμευτείτε κύριε Υπουργέ και να εγγυηθείτε ότι οι συμφωνίες με τις ε, τρίτες χώρες θα τηρούνται. Μέχρι στιγμής Συμβούλιο και Επιτροπή περί άλλα τυρβάζουν. Και υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Το Μαρόκο που δεν τηρεί τις τιμές εισόδου, ε, ούτε τις ποσοστώσεις και βέβαια απαιτήσει φυτοϊγειονομικές που είναι πολύ διαφορετικές ε, για τις τρίτε χώρες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ σημαντική ζημία για το γεωργικό τομέα. Θα ήθελα να τηρήσουμε και τα ζητήματα, να λάβουμε υπόψη μας και τα ζητήματα για τις άκρος απόμακρες περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και τα Κανάρια νησιά. Και ένα άλλο θέμα που είναι η μπανάνα, πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Γεωργία. Συζητάμε και θα συζητάμε για την μπανάνα, αλλά θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς αν θα υπάρξει δέσμευση κοινοτική στήριξη ε, της ε, μπανάνας ε, που έχουν ως αποτέλεσμα να διακινδυνεύει η δική μας παραγωγή λόγω μείωση των δασμών. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα είστε ένας υπέρμαχος ε, του τομέα της γεωργίας που και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, Υπουργό. Σε ό,τι αφορά την επιτυχία της κοινή γεωργικής ε, πολιτικής, που είναι λίγο εφημισμός αυτό που λέω, γιατί έχει μειωθεί το εισόδημα των γεωργών κατά 5%. Και σε ό,τι αφορά τι δημοσιονομικές ε, απαιτήσει ε, τη πολιτική προπολισμού, θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σα ό,τι αφορά τη διαφάνεια την, στην αγορά εργασίας. Αντί το Συμβούλιο και άλλοι να δουν πώς μπορούν να αυξήσουν ε, την δύναμη των παραγωγών, καλύτερα θα ήταν να μειώσουν τη δύναμη άλλων παραγόντων, άλλων κρίκων της αλυσίδας, όπως οι μιλιανοπολιτές ή οι ε, μεταπητές, γιατί φαίνεται να υπάρχει ένα είδος δυσπιστίας, ε, μάλλον ε, απροθυμίας να δοθεί προσοχή σε αυτούς τους κρίκους της αλυσίδας, της διατροφικής αλυσίδας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και θέματα ηθικής είναι λέξη η οποία αναφέρεται, θα πρέπει να υπάρχει και ε, δίκαιη αλυσίδα τροφίμων, αλλά θα πρέπει να είναι και οι πρόσοδοι των γεωργών δίκαιες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση αναφέρεται εις ε, το θέμα της ε, συμφωνίας με τα κράτη Μερκοσούρ που συζητήθηκε σε μία πρόσφατη συνεδρίαση ε, και πρέπει να υπάρξει μία συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά τη γεωργία. Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας για αυτές τις διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις και πόσο πιστεύει ότι θα επηρεαστεί ο γεωργικός τομέας που είναι ένας από τους βασικούς σε αυτή την ε, διαπραγμάτευση. Δεύτερον αναφέρομαι στην ε, τεχνική γενετικής παραγωγής και καλλιέργειας και ιδίως στον τομέα της Αυστρίας διότι πιστεύω ότι αν υπάρχει αυτοδιάθεση η οποία συζητάται αυτή τη στιγμή εις το Συμβούλιο και απορρέει από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τι στρατηγική θα επί στο μέλλον την αδειοδότηση για την καλλιέργεια και παραγωγή γεννητικά τροποποιημένων οργανισμών. Ευχαριστώ η γεωργική κρίση, η κυρία Ράιμερς, έχει αφήσει παντού ε, ίχνη και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συγχρηματοδότηση που είναι ένας βασικός τρόπος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε όμως ότι ε, η συγχρηματοδότηση είναι και ένα μέσο αποκλεισμού από προγράμματα. Οπότε μπορείτε να μας πει δείτε πώς θα μπορέσει η συγχρηματοδότηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να διαμορφωθεί διαφορετικά, δηλαδή ε, πώς θα μπορέσουν ε, ε, άλλοι οργανισμοί να καλύψουν το ποσοστό των περιφερειών κατά τρόπον ώστε να συνεχίσουν να χορηγούνται οι ευρωπαϊκοί πόροι.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω μία σύντομη ερώτηση για τον προϋπολογισμό. Μαζί με το Συμβούλιο πιστεύω ότι διατυπώνουμε μία πολιτική ε, και ελπίζω θα την έχουμε και γραπτός για την γεωργική μεταρρύθμιση αλλά χρειαζόμαστε χρήματα, χρήματα και καταρχήν τις συνεισφορές των κρατών μελών. Εσείς τι κάνετε. Εμείς ζητα, εσείς ζητάτε από τα κράτη να παραμείνουν στο επίπεδο της προηγουμένης περίοδου, ζητάτε να στηριχθούμε στους ίδιους πόρους Ευρωπαϊκής Ενώστησης ή πρεσβεύετε ένα τρίτο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε ε, Υπουργέ, σας χαιρετίζω όπως και το επιτελείο σας και σας εύχομαι μία ε, καλή προεδρία. Θα έπρεπε ε, να συνεργαστούμε φιλικά μεν αλλά και συνειδητά διότι από την κατάρρευση του κομμουνισμού μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη μεγάλη ιστορική δυνατότητα ήμασταν ε, απλώς ε, ένας διάδοχος του μεγάλου κεφαλαίου που διαμόρφωνε την πολιτική στην Ευρώπη. Τώρα όμως ε, δεν θα πρέπει να παρουσιάζουμε ότι όλα είναι ρόδινα διότι υπάρχει η εμπειρία των γεωργών και ε, έχουμε και τις εμπειρίες των μετακομμουνιστικών κρατών στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι υπήρχε μία απεικιοκρατία, έπρεπε να προσφέρουμε τις αγορές μας για να πάρουμε ένα μικρό ποσοστό των ε, ε, επιδοτήσεων. Τώρα λοιπόν παράγουμε ε, βιομηχανικά προϊόντα όπως ε, η παραγωγή ζαχάρεως στην Ουγγαρία και ε, πιστεύω ότι για να πετύχει η Ουγγρική Προεδρία θα πρέπει να στρέφεται γύρω από ένα βασικό άξονα και αυτό ισχύει και στα άλλα κράτη-μέλη που έζησαν στο προκομμουνιστικό παρελθόν και ε, να ε, διαμορφωθεί μια πολιτική η οποία δεν θα είναι φιλική μόνο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και προς τους γεωργούς να συμμετέχουν και αυτοί στις συζητήσεις για όλα τα θέματα όπως και για την ε, γαλακτοκομία ε, δεν είναι λοιπόν επαρκές εσείς να ακούτε τους άλλους αλλά και να υπολογίζετε τη γνώμη που ακούτε. Επίσης η νομική προστασία, ιδίως στα νέα κράτη-μέλη. Η νομική προστασία αναφέρεται και στους γεωργούς της Δυτικής Ευρώπης που ε, έχουν παραδοθεί ανεφόρων στις μεγάλες αλυσίδες ε, των ε, υπερκαταστημάτων. Δεν έχουν πλέον οι μικροί γεωργοί κανένα δικαίωμα. Εσείς πώς σκοπεύετε να λύσετε το πρόβλημα αυτό. Μετά είπατε στην αρχή ότι ο στόχος είναι να προσφέρουμε μία διατροφική ασφάλεια εις ε, το λαό ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και θα παράγονται αλλά και θα επεξεργάζονται τα τρόφιμα ή επιτόπου. Πώς πιστεύετε λοιπόν ε, ότι θα βελτιώσετε τις συνθήκες για τους Ούγγρους γεωργούς. Σε κυρίες και Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι χρειαζόμαστε ε, ισχυρή κυνηγερική πολιτική. Αυτό θα φαντάζομαι ότι είναι και ένα σλόγγαν της Προεδρίας ε, ή αναφέρεστε και σε αξίες και μηνύματα που πρέπει να περάσουμε. αλλά ε, ε, κατά την έννοια των όσων είπε η κυρία Μαγκίνες πρέπει να σκεφτούμε λίγο. Και μερικές φορές θα πρέπει να ντρεπόμαστε με αυτά που προσφέρουμε στους γεωργούς μας. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε για τις συνθήκες με, κατά τις οποίες ζουν. Όλοι, από ό,τι βλέπω, προσπαθούν να περικόψουν ε, πόρους ε, από την ε, ΚΑΠ. Άρα τι κάνουμε εδώ. Τι είδους κοινοβουλευτική επιτροπή είναι αυτή, εάν και εμείς λέμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τους πόρους ή να συμφωνήσουμε με όσα λένε οι υπόλοιποι στα άλλα θεσμικά όργανα ή ακόμα και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα το ζήτημα των οικονομικών των γεωργών μας. Τι είδους απολαβές έχουν και γιατί δεν έχουμε και κάποιους γεωργούς εδώ να μας πούν πώς ζουν. Και τότε ίσως αλλάζαμε και γνώμη. Όλοι φοβούνται να κάνουν ισχυρές παρεμβάσεις. Γιατί αλλά ξέρετε, ε, και φοβούνται και τις παρεμβάσεις γενικά. Εάν όμως δεν κάνουμε κάποια παρέμβαση στην αγορά των ε, ε, δημητριακών, τότε θα επηρεαστούν όλοι οι τομείς. Και η χειροτροφία και άλλες και άλλοι τομείς. Η παραγωγή των σιτηρών διέπεται από τις κλιματικές συνθήκες. Εάν έχουμε έναν άσχημο χειμώνα, δεν θα έχουμε καλή παραγωγή. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα θεωρούμε απολύτως λογικά και να μην παίρνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις εμείς Νταντέν και μετά ο κύριος Λαβία. Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε που η χώρα σας ε, ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την Πολωνία θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις, άλλες για την κάπε και άλλες για τις διμερείς συμφωνίες. Στις διαπραγματεύσεις ε, με το Μερκοσούρ, η εντολή της Επιτροπής είναι πρώτερη από την ε, ε, εισδοχή της χώρας σας και μερικών άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα δραχτείτε της ευκαιρίας έτσι ώστε να απαιτήσετε μια νέα εντολή η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την πραγματικότητα, τη σημερινή πραγματικότητα της γεωργίας σε μια Ευρώπη των 27. Δεύτερη ερώτηση για την ΚΑΠ. Στη μεταρρύθμιση που παρουσίασε ο Επίτροπος, έστω και αν χρησιμοποίησε τον ίδιο όρο, δηλαδή πυλώνας, οι δύο πυλώνες που προτείνει δεν έχουν καμία πλέον σχέση με τους δύο πυλώνες που γνωρίζουμε εδώ και 12 χρόνια περίπου στην κοινή γεωργική πολιτική. Ποια είναι η εκτίμησή σας όσον αφορά αυτήν την εξέλιξη της ε, φύσης, της ουσίας ε, των ε, πυλώνων. Και ένα θέμα το οποίο αφορά και το μέλλον. Έχουμε μονάχα 7% των γεωργών κάτω από τα 35 χρόνια. Δηλαδή όλοι μεγαλώνουν πιστεύετε ότι θα πρέπει να ληφθεί καλύτερα αυτή η αλλαγή των γενεών ε, στην εξέλιξη της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μεταξύ των ε, θεμάτων που σχετίζονται με την κοινή γεωργική πολιτική υπάρχουν ε, μερικά τα οποία ενδεχομένως τον περιορισμένο χρόνο ε, που είχε ο κύριος Υπουργός στη διάθεσή του για να δώσει την θέση της Προεδρίας. Ίσως λέγω δεν είχε το χρόνο για να ασχοληθεί με κάποια σημαντικά ζητήματα. Θα τροποποιήσουμε λοιπόν την κοινή γεωργική πολιτική, θα την μεταρρυθμίσουμε. Στα πλαίσια αυτά θεωρείται απαραίτητη ε, μία μεταβατική περίοδο ή μήπω θεωρείται ότι το πέρασμα στο νέο σύστημα επιδοτήσεων, οποιοδήποτε και αν αυτό, τώρα που θα εγκαταληφθεί το παλαιό ιστορικό ε, σύστημα, ε, θα πρέπει να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη σχετικά με τις μικρές εκμεταλλεύσεις, τις μικρές αγρικίες. Ο κύριος Δες είπε ότι τα 15 εκτάρια θεωρούνται μικρή, ε, μικρή εκμετάλλευση στην ε, Λιθουανία. Αλλά ξέρετε, ε, σε μία εκμετάλλευση που παράγει σιτηρά μπορεί να έχουμε 30 μέρες δουλειά το χρόνο, ενώ σε μία ε, που ασχολείται με λουλούδια ή με λαχανικά 2.500 εργάσιμες κατά κάποιο τρόπο ώρες. Ε, επομένως ε, θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε άλλα κριτήρια διαφοροποίησης των μεγάλων από τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, είπατε ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να μειωθούν οι διακυμάνσεις. Ε, σε σχέση με αυτό έχετε κάποιες προτάσεις. Αναφέρεστε σε άμεσες παρεμβάσεις στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα μονάχα το 9% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΑΠΑ αναφέρεται στην αγορά ή αναφέρεστε ε, καλύτερα σε κάποιους άμεσους ε, μηχανισμούς ε, που χρησιμοποιούνται άλλωστε ήδη σε μη ευρωπαϊκές, μάλλον μη κοινωτικές χώρες έτσι ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα των τιμών. Ο κύριος Άνιου. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτά που δεν αναφερθήκατε. Δεν αναφερθήκατε στην ε, επερχόμενη κατάργηση των συστοιχειών κλοβών ε, για τα κοτόπουλα, ε, το οποίο θα λάβει χώρα σε ένα χρόνο. Ε, θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν το αναφέρατε και ε, ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα, ε, ξέρετε ότι στη διάρκεια της Προεδρίας σας αρχίσει να εφαρμόζεται και ξέρετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά τον αριθμό των αυγών που τίθενται στην αγορά. Τι θα κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευρύτατη η συμμετοχή στην συζήτηση, αγαπητέ Υπουργέ. Δυστυχώς, Έχουμε ή μάλλον εσείς έχετε στην ε, διάθεσή σας 12-13 λεπτά γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα της ημερησία διατάξεω μέχρι τις 6. Μετά έχουμε ε, άλλο θέμα στη ημερησία διάταξη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τι ε, απαντήσεις σας και σας δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανένα ερώτημα που δεν θα ήθελα να απαντήσω. Και αν ε, δεν αναφέρθηκα σε κάποιο θέμα προηγουμένως υπάρχει κάποιος λόγος. Παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι ένα θέμα που να μην αποτελεί ένα ουσιαστικό θέμα της Ουγγρικής Προεδρίας και αυτό ε, το εξηγεί. Αλλά θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση σχετικά με τη συστοιχεία κλοβών. Δηλαδή πώς ε, αυτά τα προβλήματα συνδυάζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα εκπνεύσει η προθεσμία όσον αφορά τις συστοιχίες των κλοβών και βλέπετε ότι πολλοί δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν δηλαδή υπάρχουν ακόμη 30% οι οποίοι κρατούν τα κοτόπουλα σε συνηθισμένα κλουβιά και ενδέχεται ε, αυτό, αυτή η εξέλιξη να οδηγήσει σε ανισότητες της αγοράς και γι' αυτό έπρεπε να βρεθεί μία μέση οδό η οποία να είναι αποδεκτή από όλους. Ε, πρόκειται για επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους πτυνοτρόφους οι οποίοι Εντό εντός 10 ετών δεν είχαν καμία οικονομική δυνατότητα ή ενίσχυση για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε πιο σύγχρονα κλουβιά. Υπάρχει και μια οικονομική κρίση η οποία έπληξε αυτούς τους ορνηθοτρόφους και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει επίσης να μας απασχολήσει και εδώ και στο Συμβούλιο. Εδώ τουλάχιστον ακόμη ισχύει η νομοθεσία. Τώρα έρχομαι ε, σε άλλα θέματα. Βέβαια καλό θα ήταν να είχα και άλλο χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Εάν η πολλαπλή συμμόρφωση θα εφαρμοστεί ή όχι μετά το 2014 είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού. Και υπάρχει και ένα άλλο βασικό θέμα, δηλαδή ένα άλλο μελλοντικό θέμα, εάν ε, δηλαδή θα πρέπει ε, να συζητήσουμε ε, να υπάρχουν συγκεκριμένες ενισχύσεις για ορισμένα θέματα, δηλαδή εστιασμένες δηλαδή για την υγεία παραδείγματος χάρη και να υποφελούνται αυτοί οι οποίοι όντως εργάζονται. Ε, δηλαδή πρέπει να προβούμε σε ένα ορισμό του ενεργού παραγωγού και θα δούμε ότι πολλοί αποκλίνουν από αυτό τον ορισμό. Υπάρχουν ε, οι ε, μερικώς απασχολούμενοι, υπάρχουν γκαρσόνια που είναι συγχρόνως και παραγωγή και ε, άλλοι οι οποίοι δεν έχουν έχουν άμεση σχέση ε, με τη γεωργία αλλά αποτελούν μέρος της υπαίθρου. Και τα άτομα αυτά μέχρι στιγμής ε, στηρίχθηκαν από γεωργικές ενισχύσεις ενώ ε, τώρα έχουν προσιλωθεί στον τουρισμό και δεν είναι πλέον ενεργή παραγωγή. Θα έπρεπε κανείς να περιγράψει γράψει ακριβέστερα τους ενδιαφερόμενους για να υπάρχει πιο εστιασμένη ενίσχυση. Ε, όσον αφορά το συνολικό σύστημα των ενισχύσεων, όντως υπάρχει αιτιολογημένη ε, κριτική διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη περισσότερο ε, τα θέματα του περιβάλλοντος. Έχουμε μία εικόνα του μέλλοντος και θετική αλλά και αρνητική. Ε, και υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαν να λυθούν με απλές νομοθεσίες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο ελπίζω ότι θα είμαστε δημιουργικοί και θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να να διατυπώσουμε κείμενα τα οποία θα γίνουν αποδεκτά από τους γεωργούς ε, να υπάρξει μία προστασία του περιβάλλοντος και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Γεωργία να έχει μία μελλοντική εικόνα με μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και διατήρησή του πολλά ερωτήματα ετέθησαν σχετικά με την ονειθοτροφία, την χειροτροφία, ότι χρειάζονται μεγαλύτερες ενισχύσεις και πιστεύω ότι η τωρινή κατάσταση απέδειξε ότι ε, πρέπει να ξανασκεφτούμε και να αναθεωρήσουμε τα μέτρα αυτά στηρίξεως διότι αναλόγως των περιοχών, αναλόγως των προγραμμάτων διατίθενται τέτοιοι πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας τομέας ο οποίος θα παραβλέπεται. Όλοι θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Έχουμε πολλές διαπραγματεύσεις με τρίτα κράτη, θα μπορούσαμε με αυτό να καλύψουμε όλο το βράδυ ε, και θα μπορούσαμε συνεχώς συνεχώς να σας ενημερώνουμε για τις διεξαγόμενες ε, διαπραγματεύσεις που είναι και προς όφελος των γεωργών μας. Αλλά επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε την ε, προστασία του Ευρωπαίου γεωργού και η οικονομική κρίση βεβαίως έχει ε, και αρνητικές επιπτώσεις για τους γεωργούς. Ε, υπάρχουν και επιπτώσεις που δεν έχουν δημοσιονομική μορφή, δηλαδή ε, τα πρότυπα συμβολέων, τις προθεσμίες πληρωμής, έχουμε εισαγάγει και αυτά τα νέα στη μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και που αναφέρονται τους παραγωγούς, στους στη μεταποιητική βιομηχανία όπου υπάρχει και η ανάγκη αλλά και η ευθύνη να προταθεί ένα μεταβατικό πλαίσιο και ένα ε, μελλοντικό τελικό πλαίσιο. Βλέπω όμως ότι ο χρόνος μου περνάει. Όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση, αυτό είναι το επόμενο θέμα που θα θίξω και νομίζω ότι σε αυτήν βασίζεται το μέλλον της γεωργίας και θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιρροές των νέων κρατών μελών ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής να υπολογίσουμε και τους νέους γεωργούς γιατί χωρίς αυτούς δεν πρόκειται να υπάρξει μέλλον της γεωργίας εάν δεν αναλάβουν τη σκητάλη από τους παλαιότερους. Υπάρχουν και άλλες δηλαδή τα ταμεία τα οποία υπάρχουν ε, δεν θα επαρκέσουν και οι νέοι που ξεκινούν σε ένα επάγγελμα δεν θα ξεκινήσουν όπως ε, οι ε, προκάτοχοί τους και εδώ θα συμπεριλάβουμε και την ιδιωτική αποθήκευση. Επίσης όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα πρέπει να δούμε δούμε αν η χρηματοδότηση είναι κοινοτική ή όχι. Και πάλι το θέμα αυτό ίσως θα πρέπει να διεξαχθεί ε, και να συζητηθεί στο μέλλον. Εγώ πάντως στηρίζω τους γεωργούς και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ Σαντόρ Φαζέκας. Πραγματικά σε ευχαριστώ σου. Είμαι ευγνώμων μάλιστα για την ε, διαθεσιμότητα που έδειξες. Είμαι βεβαίως ότι ε, θα είναι μεγάλη η συμβολή της ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή και καλή τύχη σε αυτό το ξεκίνημα της Ουγγρικής Προεδρίας. Ένα λεπτό διακοπή και συνεχίζουμε με τη διοξίνη. Τελευταίο σημείο, πού πάτε, λέει ο πρόεδρος, γυρίστε στη θέση σας, καθίστε, έχουμε κι άλλα. Είναι δυνατόν να φύγει ο George Lyon, δεν γίνεται αυτό. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη τη σήμερα είναι το σκάνδαλο της διοξίνη στην Γερμανία και παρουσίαση λοιπόν της κατάστασης Καθώ επίση και αναμένω μηνύδες τη Επιτροπή από του εκπροσώπους τη Επιτροπής. Ξέρετε φαντάζομαι ότι ο Επίτροπος ε, ε, Νταλή την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και τη διάρκεια τη ε, συζήτηση στην Ολομέλη ανακοίνωσε λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο νέων μέτρων έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά ει το μέλλον θεωρήσαμε ότι πρέπει να συζητήσουμε εκ νέου το θέμα της διοξίνης εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας και θα δώσω λοιπόν αμέσως τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικό Διευθυντή της, ε, ε, ε, για θέματα υγιεινής της DG Sanko, στον κύριο Πουντλέ. Η κυρία Μαραθουέλα, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ενδεχομένως, ναι δεν ήρθε και ενδεχομένως κάποιος που θα έχει έρθει στη θέση της μπορεί να πάρει το λόγο μετά. Ο κύριος Πουντλέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ε, καλέσατε εδώ έτσι ώστε να σας περιγράψουμε λίγο πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Ε, μοιράσαμε ένα μικρό διάγραμμα, ελπίζω να το έχετε όλοι, έτσι ώστε να σας εξηγήσουμε εν συντομία την ε, κατάσταση. Γνωρίζετε ότι μια εταιρεία που κατασκευάζει ε, biodiesel έδωσε ε, πρώτη ύλη 206 ε, τόνους λίπους ε, στην εταιρεία FeedFat που ε, ανακάτεψε το λίπος αυτό με άλλο λίπος άλλης προέλευσης και με τη σειρά της η εταιρεία αυτή ε, πούλησε το λίπος σε διάφορες, 25 στον αριθμό συγκεκριμένα, εταιρείες σε διάφορα ομόσποδα κρατήδια. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν το λίπος ε, σε, ε, ε, στην, για την τροφή οτόκων ορνήθων, χείρων, χειριδίων κλπ. Contamination qui a été Γνωρίζετε ότι ο βαθμός μόλυνσης που βρέθηκε ε, στα, ε, σε αυτά τα προϊόντα, στα ζώα, ε, κυρίως δε σε το γάλα και το κρέας των ζώων που ετράφησαν με μολυσμένα, μολυσμένες ζωοτροφές δεν προκαλούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ε, τα ποσοστά βεβαίως ε, ξεπερνούν ε, τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τις αναλύσεις αλλά δεν, είναι, δεν βρίσκονται σε επίπεδο εξαιρετικά κρίσιμο. Δηλαδή τα επίπεδά τους είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που είδαμε στην κρίση της Ιρλανδίας από 2,5 χρόνια. Είναι δύο φορές παραπάνω από το ε, συγγνώμη, 200 φορές παραπάνω από το κανονικό ήταν τότε στην Ιρλανδία. Εδώ βρισκόμαστε σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα. Ας πούμε, 1,5 φορά παραπάνω ε, για το κρέας ε, και 4-5 φορές παραπάνω από το κανονικό για τα αυγά. Αυτό σημαίνει ότι η μόλυνση έχει υπάρξει, ναι, αλλά η μόλυνση αυτή δεν ε, αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η μόλυνση αυτή ε, βεβαίως καταγράφεται γιατί ξεπερνάει τα όρια τα οποία έχουμε θέσει και υπάρχει πάντα κίνδυνος μόλυνσης των ε, ανθρώπων ε, διότι ε, η κάθε, ο κάθε βαθμός μόλυνσης ε, κατά κάποιο τρόπο αποθηκεύεται στον οργανισμό και η επόμενη μόλυνση έρχεται να προσθεθεί στα επίπεδα τα οποία υπήρχαν προηγουμένως. Άρα δεν είναι δυνατόν ο καταναλωτής να καταναλώνει διαρκώς προϊόντα τα οποία είναι μολυσμένα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία τα οποία ήθελα να σας αναφέρω. Επίσης να σας πω ότι φρονούμε πως το σύστημα ειχνηλασιμότητας έτσι όπως έχει εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσε καλά, ότι η Γερμανία μέσω του συστήματος ε, γρήγορης ε, ε, ειδοποίησης ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27 Δεκεμβρίου το βράδυ έγινε η ενημέρωση από την Γερμανία. Εμείς άμεσα ενημερώσαμε τα κράτη-μέλη. ακολούθησαν καθημερινές αναφορές από πλευρά της Γερμανίας που μας κρατούσε ενήμερους για την εξέλιξη της κατάστασης. Επίσης βρισκόμαστε σε επαφή με τρίτες χώρες γιατί ε, μία ε, από τις μεγάλες μας ανησυχίες ήταν να ξέρουμε εάν ε, σφάγια ή προϊόντα προερχόμενα από τις, από τις φάρμες που, που χρησιμοποίησαν αυτές τις μολυσμένες τροφές είχαν βγει σε τρίτες χώρες. παρόλο που δεν διαπιστώθηκαν ε, εξαγωγές προς τις χώρες αυτές από τις ε, παρτίδες που μας απασχολούσαν. Παρόλα αυτά λέγω, ε, κάποιες τρίτες χώρες πήραν μέτρα κυρίως όσον αφορά την απαγόρευση εισαγωγής κυρίως χειρίου κρέατος. Η Ρωσία, ας πούμε, μπλοκάρισε εν μέρη τις εισαγωγής χειρίου κρέατος και επίσης εφήρμοσε επιπλέον ελέγχους. Υπήρξε διαρκής ροή πληροφοριών από, ανάμεσα στη Γερμανία, της, ε, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των χωρών μελών, έτσι ώστε να γίνουν γνωστές όλες οι διαδικασίες που έλαβαν χώρα. Βλέπετε ότι την 7η Ιανουαρίου του 2011 ε, μπλοκάρισαν οι γερμανικές αρχές 4.760 αγρικίες 4.760 λοιπόν αγρικίες ε, ε, σφραγίστηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να δώσουν πλέον ε, ούτε, ούτε γάλα, ούτε αυγά, ούτε κρέας στην κατανάλωση χωρίς να γίνουν πρώτεροι έλεγχοι. Πρόκειται για φάρμες οι οποίοι οι οποίες ε, ε, χρησιμοποίησαν ε, τις ζωοτροφές από αυτά τα 25 εργοστάσια, αλλά δεν ήταν μολυσμένες όλες οι ποσότητες ζωοτροφών. Παρ' όλα αυτά μπλοκάρισαν, μπλοκάρισαν οι γερμανικές αρχές όλες τις αγρικίες. Στις 24 Ιανουαρίου 2011, αλλά δεν έχουν αλλάξει, ε, ε, τα στοιχεία στις, ε, από, τις 20, από τις 24 Ιανουαρίου μέχρι τώρα 589 αγρικίες μονάχα έχουν μείνει μπλοκαρισμένες και θα απεμπλακούν μονάχα, θα απελευθερωθούν δηλαδή οι παραγωγές τους μονάχα εάν βάσει των δειγμάτων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με τους ε, Γερμανούς ε, ε, προσπαθήσαμε να δούμε πώς ξεκίνησε το πρόβλημα, γιατί αυτά τα λύπη ήταν μολυσμένα, αυτά που ξεκίνησαν από την εταιρεία παραγωγής biodiesel. Δεν έχουμε ακόμα σαφή απάντηση. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι υπήρξε λάθος ανθρώπινο. Ανθρώπινο σφάλμα λοιπόν ε, γιατί αυτό το, αυτή η μονάδα παραγωγής στο Μπέζελ της ε, Γερμανίας ε, είχε αφενός τμήμα παραγωγής λιπαντικών ουσιών για την βιομηχανία αλλά και λίπους για τις ζωοτροφές. Και ένα ενδεχόμενο λοιπόν ήταν σε αυτό το εργοστάσιο ενδεχομένως υπήρξε λάθος, σφάλμα ανθρώπινο, ε, ενδεχομένως το αποθηκευμένο λίπος το οποίο χρησιμοποιήθηκε να, ήταν, να μπήκε σε λάθος υλό. Άλλο ενδεχόμενο ε, είναι το ενδεχόμενο της απάτης, αλλά ακόμα κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Γιατί η εταιρεία αυτή ε, στο, που βρίσκεται στο Ιντερσεν Μπέζελ Ε, έλαβε πολλές, ε, πολλές παρτίδες ε, λίπους. Οι τέσσερις μονάχα, οι τέσσερις παρτίδες ήταν μολυσμένες. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι υπήρχε λάθος εάν πρόκειται για μία παρτίδα, αλλά εδώ έχουμε πολλές παρτίδες. Τέσσερις παρτίδες είναι δύσκολο να γίνει τεχνικό λάθος, ανθρώπινο λάθος, ε, σε τέσσερις παρτίδες. Ε, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, η γερμανική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει, ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Ω εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το είχε πει άλλωστε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, ο, ο Επίτροπος και το επανέλαβε χθε ε, ε, του ενώπιον των Υπουργών Γεωργία στο Συμβούλιο Γεωργία. Αποφάσισε λοιπόν ο Επίτροπος ε, να θέσει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο τεσσάρων μέτρων έτσι ώστε να αποσαφινιστεί περαιτέρω η νομοθεσία και να αποφευθούν μελλοντικά προβλήματα. Πρώτο μέτρο είναι η πιστοποίηση των ε, ε, εταιριών ε, που χειρίζονται αυτά τα λύπη. Μια πιστοποίηση η οποία θα είναι πολύ πιο αυστηρή από την απλή καταγραφή. Ε, αυτό σημαίνει ότι εάν ένα εργοστάσιο θέλει ε, να χειρίζεται λύπη, τότε θα πρέπει να ε, ελεγχθεί από μια επιτροπή η οποία θα ελέγξει τα συστήματα αυτοελέγχων, το, όλη την αλυσίδα επεξεργασίας και παραγωγής κτλ. Δεύτερο μέτρο διαχωρισμός της ροής παραγωγής σε αυτές τις εγκαταστάσεις, όταν, σε αυτά τα εργοστάσια, όταν ε, αυτές ασχολούνται ε, και με τα ε, λίπη, τις λιπαντικές ουσίες, βιομηχανικά λίπη λοιπόν, και όταν, όταν παράγουν λίπη για την κτηνοτροφία. Επίσης, φυσικός διαχωρισμός όταν σε κάποιο εργοστάσιο ε, δουλεύει κανείς και με τα δύο είδη λίπους. Όχι εάν οι εγκαταστάσεις έχουν, είναι διαφορετικές και απέχουν ε, μεταξύ τους. Επίσης, στις εγκαταστάσεις αυτές που δουλεύουν και με τα δύο είδη λίπους ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν νέα μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει διαφοροποίηση, δηλαδή να μην, ε, δηλαδή το στόμιο των σωλήνων πούμε, να έχει διαφορετική διάμετρο στη μία ή στην άλλη περίπτωση έτσι ώστε να μπορεί να αποφευχθεί ε, το ανθρώπινο λάθος. Όπως είναι ας πούμε διαφορετικό το στόμιο ε, σε, ένα, σε μία αντλία βενζίνης εάν πρόκειται για βενζίνη για καταλυτικά αυτοκίνητα ή συμβατική βενζίνη. Τρίτο μέτρο. Βελτίωση του ελέγχου των επιπέδων διοξίνης, δηλαδή ε, έλεγχη διοξίνης στα εργοστάσια τα οποία ε, χειρίζονται λύπη. Είτε πρόκειται για ε, λύπη ζωικής προέλευσης, ε, όπως ήταν η περίπτωση του προβλήματος στο Βέλγιο, είτε φυτικής προέλευσης, ε, με ελέγχους υποχρεωτικούς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι προαιρετική η έλεγχη, επομένως έλεγχη τακτική, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί ε, η περιοδικότητα των ελέγχων, αλλά έλεγχη υποχρεωτική πλέον σε όλα τα εργοστάσια τα οποία ε, ε, χειρίζονται τα λύπη. Ξέρουμε ότι έχουμε ήδη το παράδειγμα του Βελγίου που μετά από την βελγική κρίση διοξινών ε, έχει εφαρμόσει πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία, αυστηρούς κανόνες για τα λύπη ζωικής προέλευσης. Μόνο για τα λύπη ζωικής προέλευσης όμως. Και γίνεται έλεγχος για τη διοξίνη και για το PCB. Τέταρτο μέτρο. Τα εργαστήρια τα οποία κάνουν τις αναλύσεις ε, θα πρέπει να υποχρεούνται να ανακοινώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα μονάχα ε, αυτή τη στιγμή μονάχα οι εταιρείε ε, οι ίδιες οι οποίες κάνουν τον αυτοέλεγχο υποχρεούνται να αναφέρουν τα αρνητικά αποτελέσματα. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στα ιδιωτικά εργαστήρια ε, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής μηχανισμός αναφοράς, auto reporting σε εθνικό επίπεδο. Αυτά είναι λοιπόν τα τέσσερα μέτρα τα οποία τώρα μελετούμε και τα οποία συζητούμε με την βιομηχανία τροφίμων. Πρέπει να σας πω δε ότι την επόμενη εβδομάδα ε, έχουμε συνάντηση με εκπροσώπους όλων αυτών των εργοστασίων αυτής της βιομηχανίας και ευελπιστούμε ότι αρκετά σύντομα θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, αυτό το πλέγμα μέτρων. Και βεβαίως θα υποβληθεί για έλεγχο στο Κοινοβούλιο το νέο αυτό σύστημα. Ε, προσπαθούμε λοιπόν μέσω των νέων μέτρων να αποφύγουμε το ανθρώπινο λάθος και να ελαχιστοποιήσουμε το ενδεχόμενο απάτης. Κατανοείται βεβαίως ότι απάτη μηδενική δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μηδενίσουμε το ενδεχόμενο απάτης. Απλώς μέσω της αύξησης των αναλύσεων και των ελέγχων ε, είτε ε, ε, εκεί που παράγονται τα λίπη, εκεί που αναμειγνύονται με το καλαμπόκι ή με τη σόγια. Εκεί υπάρχει πάντα περίπτωση απάτης λόγω της τιμής, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να ελοχιστοποιήσουμε την απάτη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν βρισκόμαστε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποκλέ. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, πρέπει να εγκαταλείψουμε την αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα δώσω το λόγο μονάχα ε, σε δύο-τρεις ε, συναδέλφους που έχουν εγγραφεί και δυστυχώς θα πρέπει να συνεχίσουμε αύριο μετά από τη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον κύριο Ρώσου, Χόσλινγκ. και μετά Δανέλης. Αυτά. και η κυρία Γέγκλε μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή. Έχω πολλά θέματα τα οποία θα ήθελα να διευκρινίσω και θα θέσω μόνο ελάχιστα λόγω χρονικού περιορισμού. Διότι ε, εχθές παρουσιάστηκε το πρόγραμμα στην ε, Γερμανίδα Υπουργό για να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής ασφαλών ζωοτροφών ε, τα ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι γεωργοί περιμένουν να κάνουμε τα πάντα κατά τρόπον ώστε και στις 27 χώρες να υπάρχει ένα, έγγραφο, ένα επαρκές επίπεδο ε, χεγγίων. αλλά αυτό θα πρέπει να ε, αποβεί πολύ δύσκολο και αυτό ήδη το διεπίστωσαν οι Γερμανοί γεωργοί διότι διαπιστώσαμε ότι το κρέας και τα αυγά ήταν καθαρά παρόλα αυτά όμως έκλεισαν τα σύνορά τους η Ρωσία ε, και ε, ε, περαιτέρω επιπτώσεις απεφεύθησαν την τελευταία στιγμή. Χρειάστηκε να πέσουν οι τιμές τραγικά και να χαρίσουμε τα προϊόντα. Οπότε θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επέτρεψαν αυτό το πρόβλημα. Διότι υπάρχει μία αποσταθεροποίηση των καταναλωτών. Οι γεωργοί έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες ε, και ε, ε, λόγω αυτών των εγκληματικών πράξεων περίπου 600 γεωργοί υφίστανται αυτές τις επιπτώσεις και πρέπει να εγκαταλείψουν τις επιχειρήσεις τους. Στην τωρινή συζήτηση μιλάμε για την ευθύνη και την εξασφάλιση αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ασφαλιστής ο οποίος πρόκειται να καλύψει αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα μιλάμε για ζημιές 100 εκατομμυρίων ευρώ ίσως και παραπάνω άρα χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό ταμείο όπου θα πληρώνει η διατροφική βιομηχανία της Ευρώπης και θα καλύπτει αυτά τα ποσά. Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει ορισμένα σημεία του προγράμματος δράσεώς μας και που δεν θα επαναλάβω τώρα λόγω έλλειψης χρόνου. Αλλά ε, ε, μέχρι στιγμής ε, δεν υπήρχε τέτοια εμπλοκή των ιδιωτικών εργαστηρίων δικαστηρίων. Ειδοποιούσε για τα αρνητικά αποτελέσματα κανείς ε, τους, την επιχείρηση και όχι ε, ε, το κράτος. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω μέχρι πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιμένει για να καταστήσει πιο αυστηρή την νομοθεσία της ιδίως για άλλα θέματα και όχι μόνο για την διοξίνη διότι ότι ε, ο Υπουργός μας είπε ότι θα υπάρξει μια επιτροπή που θα έρθει, μια, ε, θα έρθει στη Γερμανία εντός των επομένων ημερών ε, για να εξετάσει την κατάσταση. Θα ήθελα να ξέρω ποιες θα είναι οι εντολές που θα έχει αυτή η αντιπροσωπεία. Με εκπλήσει ο κύριος Χόισλινγκ. Με εκπλήσει που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να υπάρξει αναδρομική εποπτεία διότι πιστεύω ότι το σύστημα του αυτοελέγχου δεν ε, ε, πρέπει απλώς να υπάρχει αλλά να ε, ενισχυθεί διότι μέχρι στιγμής σε τέτοια ευαίσθητα τρόφιμα ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αρχές και τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να επιληθεί το θέμα αυτό θετικά, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια διότι ορισμένες επιχειρήσεις απλώς ε, ε, ε, δήλωσαν ότι χρεοκόπησαν και τράβηξαν την ουρά τους από το παιχνίδι. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς θα λειτουργήσει το θέμα στο μέλλον. Θα υπάρχει μία δοκιμή για να δούμε αν κάποιος είναι κατάλληλος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν κατάλαβα ακριβώς πόσο θα ελέγχει κανείς την επεξεργασία σε διάφορες επιχειρήσεις αν η μία κάνει ζωοτροφές και η άλλη ε, κάνει τρόφιμα. Ε, επίσης ε, μπορείτε να μας πείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσες δοκιμασίες θα πρέπει να γίνονται και πού στην Ευρώπη διότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ δαπανηρά. Μιλήσατε για 200 τόνους. Δηλαδή πού βασίζεται το όριο αυτών των 200 τόνων εγώ δεν καταλαβαίνω. Ευχαριστώ κύριος Δανέλης και μετά η κυρία Ρέιμερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αντιθέτως από την ε, προσπάθεια υποβάθμισης και εφησυχασμού αλλά και την ε, αυτάρεσκη διαπίστωση ότι το σύστημα λειτουργήσε ικανοποιητικά την περασμένη εβδομάδα από το στόμα του Επιτρόπου και σήμερα από τον ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής Νομίζω ότι αυτή τη φορά το, το, σκάνδαλο με τις ε, ε, διοξίνες στις ζωοτροφές είναι πολύ σοβαρότερο γιατί έχει σοβαρότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από οποιοδήποτε στο παρελθόν. Πρώτα απ' όλα εξελίσσεται σε μια χώρα όπως η Γερμανία, όπου είναι γνωστή η παράδοση πειθαρχία στη χώρα αυτή, καθώς επίσης και η αξιόπιστη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου. Αν αυτό λοιπόν συνέβη στη Γερμανία, φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπου ο καθένας προσπαθεί να αυξήσει τα κέρδη του μειώνοντας τα κόστη, παρουσιάζεται ακόμα πιο ανίσχυρο το σύστημα το οποίο ακολουθούμε ελέγχου μέχρι σήμερα, το οποίο φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί σημαντικά σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτο, πόσοι έλεγχοι γίνονται αξιόπιστοι, παίρνοντα υπόψη τα κόστη βεβαίω των ελέγχων αυτών. Και δεύτερο, ακολουθείται ο έλεγχο από τι σοβαρότητα μέτρα χειρώσει, Γιατί αν δεν υπολογίζει ο όποιο επιχειρηματία ε, ε τη διαφορά κέρδου από το τι θα κληθεί να καταβάλει σε περίπτωση που συλληφθεί να παρανομεί, βεβαίω δεν δεν θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ απλούστατα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να πω ότι αν υπάρχουν ποινικέ ενέργειες ακόμη και οι πιο σκληροί έλεγχοι δεν θα τις αποφύγουν αλλά μια πολύ απλή λύση θα ήταν να χρωματίζει κανείς τις ε, ουσίες ελέγχου για να βλέπει κανείς τι υπάρχει μέσα στο περιεχόμενο. Ευχαριστώ κυρία Ρέιμερς, ε, κυρία Γέγκλε και μετά ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω επίσης να είμαι ε, σύντομη ενώ θα μπορούσαν πολλού να πούμε. Δεν ήξερα ότι αυτό θα το ξαναβίωνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έζησα μία φορά και φτάνει. Το γεγονός ότι τώρα συμβαίνει στη Γερμανία είναι επιπλέον επιβάρυνση διότι λέγαμε πάντοτε ότι κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Εάν υπάρχει όμως μία εγκληματική ενέργεια, ό,τι και να κάνουμε δεν θα την αποφύγουμε. Απαιτώ λοιπόν δύο πράγματα. Ο καταρχήν η Γερμανία να απαντήσει αμέσως με σαφείς και αυστηρές κυρώσεις. Εάν μιλάτε για την πτώχευση θα μπορούσαμε ε, να το έχουμε λύσει νομοθετικά στο παρελθόν. Επίσης δεν είναι δυνατόν ε, η διατροφική βιομηχανία να ανθεί και να πλήττονται οι ε, Και πρέπει να βρεθεί ένα σωστό δρόμος πέραν των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή η υγιεινή για τις ε, ζωοτροφές και το, η σχετική οδηγία πρέπει να αναθεωρηθούν για να μην διαχωρίζει μόνο κανείς τα βιομηχανικά λύπη από τα, φυτικά, τα, ζωικά λύπη αλλά για το πόσο διεξάγεται η μεταφορά και να δούμε τις, ε, τους αριθμούς των ε, λοιπόν που εισάγονται στη Γερμανία διότι δεν επιτρέπονται τα ζωικά λύπη. Μακροπρόθεσμα λοιπόν χρειάζεται ε, μία ε, σωστή και σοφή ε, πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γιάρ και μετά ο κύριος Σεκερέσκη και έτσι θα κλείσουμε. Ναι, ε, το, το θέμα είναι θέμα ελέγχων. Ό, όντως θα πρέπει να διαπιστώσουμε πού γίνονται τα περισσότερα λάθη. Και ε, Βεβαίω θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο και τους ε, κανόνες, αλλά να μην βαραίνουμε διαρκώς ε, τους κανόνες, να δούμε πού γίνονται τα λάθη, γιατί τελικά το λογαριασμό τον πληρώνουν οι γεωργοί. Αυτοί έχουν όλο και περισσότερα προβλήματα. Άνιου, θέλετε να πείτε κάτι. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε επιπλέον ε, ε, κανονισμούς. Έχουμε τρεις κανονισμούς και μία οδηγία. Δεν θέλουμε άλλη νομοθεσία. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τρία συστήματα ασφάλειας στην αλυσίδα και νομίζω ότι πλέον τα, τα θα πρέπει το καθένα χωριστά να βάλουν επιπλέον θέματα. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από την Επιτροπή. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να εγκαταλείψουμε την αίθουσα. Δεν ξέρω εάν μπορείτε ε, στην γραμματεία να αποστείλετε γραπτά απάντηση στα τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα συναντηθούμε αύριο στις 9.30. 9 οι συντονιστές, 9.30 η ε, Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Wow, wow. What time is it?